Αγαπητές φίλες και φίλοι, αρχίζουμε τη δημόσια ακρόαση σχετικά με το ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών ραδιοτηλεπτικών μέσων. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες, οι οποίοι όλοι έχουν θητεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα της ραδιοτηλεόρασης, της οικονομίας, της κοινωνίας, της τεχνολογίας σε αυτό το τομέα. Και πριν περάσω στο πρόγραμμα, θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσουν και τη βάση της συζήτησης και του προβληματισμού των οποίων έχουμε να παρουσιάσουμε σαν Επιτροπή Πολιτισμού. Καταρχήν, θα ήθελα επιγραμματικά να πω ότι ο τομέας των δημόσιων οπτικοακουστικών αποτελεί μια υπηρεσία γενικού συμφέροντος. Ορισμός της αποστολής τους εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα η οποία προσδιορίζει το ρόλο και τις υποχρεώσεις τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, οι δημόσιοι οπτικοακουστικοί πάροχοι είναι αποδέκτες είτε μιας κρατικής οικονομικής ε, ενίσχυσης άμεσης είτε έμεσης μέσω των υποχρεωτικών εισφορών ή τελών που καταβάλλονται από το ίδιο το κοινό, από τους ίδιους τους πολίτες. Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των κρατών μελών αποσαφηνίζεται στο συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συνθήκης σχετικά με το σύστημα της δημόσιας τηλεόρασης στα κράτη-μέλη. Η βασική διαφοροποίηση των δημόσιων μέσων είναι ότι η παροχή των δημόσιων υπηρεσιών εκ μέρους τους δεν ανταποκρίνεται μόνο σε εμπορικά κριτήρια και στην εξασφάλιση των πλέον δημοφιλών προγραμμάτων με στόχο την επίτευξη υψηλής τηλεθέασης, αλλά κυρίως στο κριτήριο εξασφάλισης μιας έγκυρης και αντικειμενικής ενημέρωσης. Υπάρχει το στοιχείο της ποιότητας και αυτό το βλέπουμε σε πολλές εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι όμως γεγονός αναμφισβήτητο ότι η δημόσια τηλεόραση δεν αποτελεί μια παραδοσιακή υπηρεσία οικονομικού ε, γενικού ε, συμφέροντος της αγοράς, αλλά έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύω ότι και οι συγητές, οι εμπειρογνώμονες θα μας τα αναφέρουν σχετικά με τις παραδοσιακές δημόσιες, ε, υπηρεσίες. Μία πολύ μεγάλη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν ο δημόσιος τομέας είναι αυτή της τεχνολογικής επανάστασης όπου οι πλατφόρμες διανομής, τα μέσα διείσδυσης μόνο πολλαπλασιάστηκαν με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ψηφιακή τηλεόραση αλλά και την μοντέρνα κινητή τηλεφωνία που έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό σε επίπεδο αγοράς. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, σήμερα καλούμαστε να εξετάσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο και τη λειτουργία που συνεχίζει ε, να εκπληρώνει η δημόσια τηλεόραση σε αυξημένες συνθήκες και απαιτήσει της αγοράς. Καλούμαστε σήμερα να απαντήσουμε μεταξύ των άλλων σε ορισμένα βασικά ερωτήματα σχετικά με το ψηφιακό μέρισμα και την κατανομή των σημαντικών συχνοτήτων που απελευθερώνονται, πώς μπορεί να διασφαλιστεί η δημόσια ραδιοτηλεόραση ότι θα έχει ισότιμη πρόσβαση, ποια είναι η ισορροπία που θα πρέπει να επιτευχθεί ανάμεσα στην ανάγκη αφενός για άνοιγμα των ραδιοσυχνοτήτων σε νέους φορείς που παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες και την ανάγκη διασφάλισης του πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων. Κατά πόσο και σε ποιο βαθμό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον οφείλει να έχει επίδραση στο περιεχόμενο των υπηρεσιών της ραδιοτηλεόρασης σε ποιο βαθμό και κατά πόσο διασφαλίζεται ο έγκυρος ρόλος και σκοπός για την ενημέρωση και ποιοτική ψυχολογία. Ως προς τη χρηματοδότηση, η Επιτροπή έχει βγάλει ένα σχέδιο ε, ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Κατά πόσο απαιτείται επαναπροσδιορισμός των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών και προς ποια κατεύθυνση. Τέλος, πώς θα διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των δημόσιων παρόχων οικονομικά και θεσμικά στο νέο οικονομικό, τεχνικό και κοινωνικό περιβάλλον το οποίο αναπτύσσεται. Με βάση έναν μικρό εισαγωγικό θα ήθελα να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας και όπως βλέπετε στο πρόγραμμα έχουμε χωρίσει την ακρόαση σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά το ρόλο της δημόσιας, των δημόσιων οπτικοακουστικών στη, ε, και ε, θα ήθελα να περάσω αμέσως ε, να δώσω το λόγο στον κύριο Πέρε Οριόλ Κώστα από το Πανεπιστήμιο ε, ε, της Βαρκελόνης, ε, University Professor of Political Communication, University Autonom de Barcelona και θα ήθελα να τονίσω ότι ο χρόνος είναι 10 λεπτά έτσι ώστε για να έχουμε επαρκή χρόνο για ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Κώστα, έχετε το, ρόλο, το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας απευθύνω ε, χαιρετισμού εκ μέρους των εμπειρογνωμόνων. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μου θα σας μιλήσω για τον ε, απαρίθμηση πέντε μεταβλητών για να μπορέσουμε να καθορίσουμε το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης στο παρόν οπτικοακουστικό σύστημα πρώτη μεταβλητή. Οι μεγάλες ε, δυσκολίες που έχουν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί να προσφέρουν προγράμματα ποιότητας. Η ιδιωτική τηλεόραση δεν δίνει στην κοινωνία αυτά τα οποία τη ζητάει η κοινωνία και θεωρείται πολλές ε, φορές ε, σαν κλισέ αυτό που λέω, σαν κοινοτυπία. Αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχει πρόβλημα στην ε, προσφορά των ιδιωτικών τηλεοπτικών καλενιών. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όλο και περισσότερο εξελίσσονται τα δημόσια κανάλια με πρακτικές πολύ διαφορετικές από αυτό του κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζουν τα κρατικά κανάλια. Φερρυπίν, πώς εξελίσσονται οι ειδήσει. Στις ειδήσει των ιδιωτικών καναλιών έχουμε πολύ σύντομες ειδήσει, η μεν καμία σχέση με τις δε και πολλές φορές ε, σχεδόν κίτρινου περιεχομένου. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναφέρουμε και κάποια άλλα στοιχεία. Στην χώρα μου τουλάχιστον πολλές φορές ε, καλούνται από τα ιδιωτικά κανάλια ε, διάφοροι άνθρωποι που είναι λίγο εγκληματίε ή λίγο παράνομοι εν τους πληρώνουν για να εξηγήσουν τι κάνουν στη ζωή του και πώς ζουν. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όλο και περισσότερο βλέπουμε να <laughs> ακολουθούνται πρακτικές που έχουν σχέση λίγο με τις ειδήσει και λίγο με κάποια reality προγράμματα ή προγράμματα στα οποία έχουμε συμμετέχοντες στους οποίους έχει δοθεί χρήμα για να συμμετάσχουν και για να διανθίσουν το πρόγραμμα. Βλέπετε λοιπόν το και περισσότερο απομακρύνουν το κοινωνικό τους ρόλο τα ιδιωτικά κανάλια. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο δεύτερο σημείο. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο λοιπόν να βρεθεί μια τα σταθερή ε, βάση στην οποία να συζητήσουμε τις, ε, τα κρατικά κανάλια, τα δημόσια κανάλια. Για να εξηγήσω, το λέω αυτό για να εξηγήσω το εξή. Πολλοί παρακολουθούν τα κρατικά κανάλια, αλλά συγχρόνω κριτικάρουν. Λέγουν πολύ λίγοι τα βλέπουν αυτά τα κανάλια. Και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, αρχή της επικουρικότητας. Εδώ δεν μπορεί να παρέμβει όπως παρεμβαίνει στα ιδιωτικά κανάλια το κράτος. Πολλές φορές βλέπουμε ότι για κάποια προβλήματα φταίει η αρχή της επικουρικότητας. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί αυτή η δημόσια κρατική υπηρεσία, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει δουλειά. Και ξέρουμε ότι εσείς στο Κοινοβούλιο ασχολείστε με αυτά τα θέματα, με θέματα τα οποία μπορεί να προσφέρει ο δημόσιος τομέας τηλεόραση. Θα ήθελα να μιλήσω για την, ε, αυτό το οποίο Εσείς ονομάζετε ψηφιακός ε, αλφαβητισμός, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο βοηθά τη δημόσια τηλεόραση να βελτιώσει την εικόνα της, διότι ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της κρατικής τηλεόρασης. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα είδος, πρέπει να κινηθεί στην επικουρικότητα η δημόσια τηλεόραση και πρέπει να βελτιωθεί η εικόνα της δημόσιας τηλεόρασης που με τη σειρά των ετών έχει κάπως αμαυρωθεί θα έλεγα, έχει μειωθεί. Μετά ο ρόλο της ε, ε, δημόσιας τηλεόραση έναντι της τεχνολογίας και των εξελίξεων στην τεχνολογία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Εάν το εξετάσουμε το θέμα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα την παραγωγή οι ε, δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα θα πρέπει να ε, παράγουν όσο δυνατόν περισσότερα δικά τους έργα και να συμμετέχουν στην παραγωγή και να παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε τοπικό επίπεδο, ούτω ώστε να αναπτυχθεί η οπτικοακουστική βιομηχανία, ο οπτικοακουστικός τομέας. Θα έπρεπε επίσης να ενθαρρύνουν νέες μορφές δημοσιογραφίας, όπως είναι η δημοσιογραφία των πολιτών, ε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το πετύχει η δημόσια τηλεόραση με τη νέα τεχνολογία, να βρει νέους τρόπους έκφρασης. Νομίζω ότι εδώ οι δημόσιοι πάροχοι μπορούν να καινοτομήσουν και μπορούν να πειραματιστούν πάνω σε αυτά και να επιτύχουν. Αυτό για την παραγωγή. Όσον αφορά τη διανομή, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η δημόσια τηλεόραση να χρησιμοποιήσει όλε τι δυνατότητε που τη δίδονται ώστε οι παραγωγές της να φτάσουν στον κάθε πολίτη. Και νομίζω ότι η σχετική οδηγία πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Η κοινή γνώμη ζητά και νέα προγράμματα και νέα ε, από τα κρατικά κανάλια, νέες θεματικές και βεβαίως πρέπει να λάβουμε και τις εξελίσσεις που αφορούν την ε, κινητή τηλεόραση. Επίσης, αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι η ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα για τον καθένα που είναι σημαντική όχι μόνο για να μπορεί να βλέπει τόσο προγράμματα, αλλά για να ενημερώνεται, όπως ενημερώνεται και από άλλες ψηφιακές δημοσιεύσεις. Τέταρτο σημείο η ανάγκη η δημόσια υπηρεσία να μην παρεκκλίνει από το στόχο του. Για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να συνδυάσει το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο, με το οποίο εσείς ασχολείστε καθώς και με τις ρυθμίσεις που γίνονται από κάθε κράτος μέλος. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες λειτουργίες της δημόσιας υπηρεσίας που δεν θα πρέπει να ξεχνούμε. Μία πολύ παραδοσιακή είναι η ανάγκη πάντα η τηλεόραση αν θέλετε ή τα μέσα να είναι ανεξάρτητα από την ε, εκτελεστική αρχή κάθε χώρας, από την εκτελεστική εξουσία. Ξέρουμε ότι ε, η πρόσβαση στον πλουραλισμό, η αποκέντρωση, η δυνατότητα να προωθηθούν και από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ε, τοπικές ε, γλώσσες, διάλεκτοι και κουλτούρες, χωρίς κανένα περιορισμό, είναι κάτι το πολύ θετικό. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι πάντα υπάρχει ανταγωνισμός των, των ιδιωτικών καναλιών. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί διότι η κρατική τηλεόραση, η δημόσια τηλεόραση πολλές φορές αποτελεί αντικείμενο ε, κρίσεων. Τώρα, Τελευταίο μου σημείο. Από οικονομικής πλευράς θα πρέπει να είναι αυτές οι δημόσιες, η δημόσια υπηρεσία της τηλεόρασης υπεύθυνη. Τι εννοώ. Ότι θα πρέπει να χειρίζονται τα κονδύλια με σωστό τρόπο. Και θα πρέπει να ακολουθούν διάφορα μοντέλα χρηματοδότησης Δηλαδή, ή ε, την χρηματοδότηση με ε, διαφήμιση ή χωρίς διαφήμιση ή να μπορεί να είναι η τηλεόραση ανταγωνιστική με την βοήθεια της τηλεόρασης, αλλά νομίζω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να, ερευνήσουμε τη δυνατότητα κάποιες ε, τηλεοράσεις να λειτουργούν με ένα μεικτό σύστημα. Δηλαδή, να μην προβάλλουν διαφημίσεις κάποιες συγκεκριμένες ώρες και κάποιες άλλες ώρες να ψυχα... ώρες δηλαδή στην οποία ε, προβάλλονται ψυχαγωγικά προγράμματα να χρησιμοποιούν τη διαφήμιση ως ε, ε, οικονομικό πόρο. Τώρα, από πού προέρχονται τα κονδύλια τα οποία θα τηλεοράσεις από φόρους ε, κρατικούς, από την ε, ε, παράδοση, από τα τέλη ραδιοφωνίας, ραδιοτηλεόρασης, από την άμεση διαφήμιση. Αυτή είναι η οικονομική πόρη των διαφόρων κρατικών τηλεοράσεων. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, η δημόσια τηλεόραση κάποιες ώρες πλέον δεν προβάλλει διαφημίσεις. Και ένα μέρος των ε, δαπανών που απορρέουν από την ε, μη προβολή διαφημίσεων καλύπτονται από κάποιο άλλο ταμείο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια ρύθμιση αλλά οποιαδήποτε ρύθμιση που αφορά τα οικονομικά θα πρέπει να γίνει με απόλυτη σαφήνεια για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Από όλα αυτά τα οποία σας είπα πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει να λειτουργεί η δημόσια υπηρεσία δεδομένου ότι παρέχει υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος. Δεύτερον, η αρχή επικουρικότητας όπως σας είπα για μένα είναι σημαντική. Τρίτον, τα προγράμματα ψηφιακής ενημέρωσης δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στο ίντερνετ αλλά να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά, νέα παιδιά όπως αυτά τα οποία βλέπω εγώ στο δικό μου πανεπιστήμιο τα οποία πραγματικά πρέπει να πω ότι αν μου επιτρέπετε την έκφραση μισούν την κρατική τηλεόραση. Πρέπει κάτι να κάνουμε για να τους φέρουμε προς την κρατική τηλεόραση, προς τη δημόσια τηλεόραση δίνοντας μια καλύτερη ε, εικόνα. Και επίσης, όπως σας είπα, σε θέματα οικονομικά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ε, σαφείς και να έχουμε μία τηλεόραση η οποία κατά την άποψή μου με το καλύτερο σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει είναι αυτό το μεικτό σύστημα. Δηλαδή ε, χρηματοδότηση εν μέρη από διαφημίσεις και χρηματοδότηση από άλλους πόρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πιέρο Ριολ Κώστα και πραγματικά το θέμα της ε, χρηματοδότησης και του τρόπου διαχείρισης των δημόσιων πόρων από την ε, κρατική τηλεόραση νομίζω ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ε, θα ήθελα να περάσω τώρα στον κύριο Ολιβιέ Ζαπιό, ο οποίος είναι General Director of, en français conseiller supérieur d'audiovisuel en France. Για 10 λεπτά, παρακαλώ, for 10 minutes. Merci, Madame le Président. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι εδώ ο συνάδελφος για οικογενικούς λόγους, τον αντικαθιστώ εγώ ο κύριος Μισελ Μπογιάν. Είπατε εσείς, κυρία Πρόεδρε, ότι η κρατική τηλεόραση είναι μία ε, υπηρεσία ε, δημοσίου ε, συμφέροντος για όλους. Βεβαίως, η δημόσια τηλεόραση ως δημόσια επιχείρηση, όπως ξέρετε, υπόκειται σε κρατική και κοινοτική οικονομική ενίσχυση και πρέπει να δούμε ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της δημόσιας υπηρεσίας. Το θέμα της δική μας ακρόσης είναι τριπλά επίκαιρο. Όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε πρώτα απ' όλα, θα γίνει αναφέρουσα ανακοίνηση της Επιτροπής για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες και τους κανόνες που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις. Δεύτερον, η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στην αγορά των διαφημίσεων, κάτι το οποίο έχει σχέση και με τις ιδιωτικές, τα ιδιωτικά και με τα κρατικά κανάλια. Και τρίτον, κάτι το οποίο είναι επίκαιρο, αν θέλετε, στο γαλλικό πανόραμα, η δημοσίευση στο τέλος της εβδομάδας μιας, ε, ενός νέου νόμου που αφορά τα δημόσια οπτικοακουστικά μέτρα. Θα σας πω λίγα λόγια κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μου και είμαι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης εάν θέλετε να μου επιβάλλετε συμπληρωματικές ερωτήσεις. Θα αναφέρω λοιπόν στον χρόνο που μου έχει δοθεί τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα, πρώτο σημείο. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες και οι περιορισμοί της κατοικής τηλεόρασης που αιτιολογούν κρατική χρηματοδότηση. Δεύτερον, γιατί θα πρέπει να, αποτελεί παράδειγμα και να μην είναι μέσα σε στεχανά αυτή η δημόσια υπηρεσία σε σχέση με τα ειδικά κανάλια. Τρίτον, γιατί αυτή η δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να στραφεί προς το μέλλον και τις νέες τεχνολογίες. Πρώτο θέμα ιδιαιτερότητα και περιορισμοί αυτής της ε, δημόσιας υπηρεσίας που αιτιολογεί κρατική χρηματοδότηση. Στη Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες, όλες οι εκπομπές δημόσιας υπηρεσίας καθορίζονται από την ε, ε, σχετική νομοθεσία και συμβάσεις που υπάρχουν μεταξύ της κάθε κυβέρνηση και τη κρατική τηλεόραση. Ποιε είναι αυτέ οι εκπομπέ. Οι εκπομπέ αυτέ με την, την έννοια είναι φερρυπίν, η αναμετάδοση των συζητήσεων τη Βουλή, διαφόρων ε, εκπομπών ε, δημοσίου ενδιαφέροντες, προεκλογικές εκστρατείες, ε, παρουσίαση υποψηφίων, αναμετάδοση Τη λειτουργία, την Κυριακή. Αυτέ είναι όλε οι εκπομπέ. αλλά ο προγραμματισμό θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτός των ιδιωτικών καναλιών, διότι υπάρχουν κάποιες απαιτήσει εκ μέρους του κοινού περισσότερες απαιτήσει από αυτές τις οποίες θα μπορούσε να έχει κανείς από, το, από ε, κάθε ιδιωτικό κανάλι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας υποχρεώνει να έχουμε ε, μουσικές ε, εκπομπές, εκπομπές ε, λογοτεχνικού περιεχομένου, αναμετάδοση κοντσέρτων, όπερας, ε, γαλλικές ε, ε, εκπομπές, ιστορικού περιεχομένου, πολιτιστικού περιεχομένου εκπομπές, γαλλικές, γαλλικού περιεχομένου αν θέλετε. Ίσως θα έπρεπε να γίνει και ένας πίνακας αξιολόγησης της κάθε εκπομπής για να δούμε πώς αιτιολογείται η παρουσία κάποιων εκπομπών και η αναμετάδοσή τους από τα κρατικά κανάλια. Υπάρχει στην Αγγλία ένα τέτοιο evaluation test, στη Γερμανία επίσης, διότι υπάρχει η ανάγκη και η βούληση να μπορεί κανείς με αντικειμενικό τρόπο να κρίνει κατά πόσον δικαιολογείται αυτή η ιδιαιτερότητα της κρατικής, της δημόσιας υπηρεσίας. Και σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, στην ε, France Television η Γαλλία επιβάλλει να σέβεται τους κανόνες της ανταγωνιστικότητας ώστε να μην στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός εκ μέρους της κρατικής τηλεόρασης. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι στα πλαίσια της αναθεώρησης οδηγίας πιστεύουμε ότι θα πρέπει επίση η Επιτροπή να σεβαστεί την αρχή της επικουρικότητας έτσι όπως προβλέπεται και να εμπιστευτεί τα κράτη ότι θα μπορέσουν να τηρήσουν αυτή την ε, βασική αρχή της υγιούς ανταγωνιστικότητα μεταξύ Δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανέφερε και ο κύριος Κώστα και ανέφερε και τη δική μας ιδιαιτερότητα. Από την 5η Ιανουαρίου στη Γαλλία έχουμε ένα μεικτό σύστημα. Δηλαδή, από κάποια ώρα και μετά, στα κρατικά κανάλια απαγορεύεται η διαφήμιση μεταξύ 8 το βράδυ και 6 το πρωί. Και στο 11 προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση διαφήμιση. Αυτό είναι ένας μεγάλος περιορισμός για την κρατική τηλεόραση. Συγχρόνως όμως είναι και η ευκαιρία να διαφοροποιηθεί η κρατική τηλεόραση από τη δημόσια τηλεόραση και να ε, μπορέσει έτσι και διάφορους περιορισμούς που υφίσταται να τους ε, αποτινάξει. Διότι πολλές φορές για να ικανοποιήσει αυτούς οι οποίοι χρηματοδοτούν τη διαφήμιση, η κρατική τηλεόραση χρειάζεται να ε, κάνει κάποιες υποχωρήσεις, τις οποίες σιγά σιγά θα ε, μπορέσει να σταματήσει. Φτάνω τώρα στο δεύτερο μέλος. Θα πρέπει η δημόσια υπηρεσία, όπως είπα, να είναι υποδειγματική και να προσπαθεί να ενώσει αντί να χωρίσει. Δηλαδή, οι δημόσιες, τα δημόσια κανάλια θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά, αν θέλετε, σε σχέση με τα ιδιωτικά και θα πρέπει τα προγράμματα τους να είναι διαφορετικά από αυτά της ιδιωτικής τηλεόρασης. Δηλαδή, για τη Γαλλία, όχι αμερικάνικα σύριαλ, ε, στα αθλητικά ε, διαφορετικού περιεχομένου εκπομπές. Η βούλησή μας όμως είναι να μπορούν οι πολύ σημαντικές, τα πολύ σημαντικά κρατικά κανάλια, το Antenne 2 και το ff στη Γαλλία, να είναι κανάλια, εάν θέλετε, δημοφιλή για όλους, που να το παρακολουθούν όλοι και όχι να γίνουν ελιτίστικα κανάλια, να μην θεωρηθούν. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει ένας πολύ καλός προγραμματισμός ώστε να υπάρχουν και κάποια προγράμματα τα οποία ο καθένας μπορεί να δει και κάποια άλλα τα οποία απευθύνονται σε κοινό ίσως πιο ε, διαφορετικό. Προβλέπετε λοιπόν στο μέλλον ε, τέτοιου είδους ε, αλλαγή στα προγράμματα ώστε να ικανοποιούνται οι πάντες, ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ απαιτητικών προγραμμάτων, αν θέλετε, που να αιτιολογούν την ιδιαιτερότητα του ε, κρατικού καναλιού και άλλα πιο γενικού περιεχομένου προγράμματα, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι πάντες. Αυτό το οποίο ξέρω ότι σας απασχολεί εσάς και την Κομισιό, είναι να μπορεί η δημόσια υπηρεσία να στραφεί στο μέλλον και κυρίως στα πλαίσια της ε, ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό θα γίνει πρώτα απ' όλα με την ε, γενίκευση του ψηφιακού συστήματος για όλα τα κανάλια της τηλεόρασης. Δεύτερον, με τις νέες ε, γραμμικές υπηρεσίες με την ε, προσωπική φορητή τηλεφωνία και εδώ η δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτές τεχνολογίες για να μην περιθωριοποιηθεί σε σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια. Τρίτος άξονας που είναι αν θέλετε και το αντικείμενο μιας νέας δημιουργίας είναι διάφορες ε, ε, υπηρεσίες online όχι γενικέ για όλου, αλλά οι οποίε επίση μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένα στη αιτήση του. Και βεβαίω εδώ ο ανταγωνισμό θα πρέπει να είναι υγιής και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα αλλά πιστεύω ότι οι δημόσιες τηλεοράσεις θα πρέπει να στραφούν ε, σε αυτή την ε, νέα τεχνολογία, την μη γραμμική ε, τεχνολογία για να μπορέσουν να ε, μην περιθωποιηθούν. Τελειώνοντας, λέω ότι σαφώς όλοι ξέρουμε ότι δεν θα πρέπει να στρεβλώσει το, η κρατική τηλεόραση τον ε, ανταγωνισμό ή αντιθέτως ε, όλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να σέβονται τους κανόνες. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να γίνει ένα ελιτίστικο κανάλι και μια ελιτίστικη υπηρεσία, αλλά μια υπηρεσία ανοιχτή σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ολιβιέ Ζαπιού. Ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι το περιεχόμενο της ε, δημόσιας τηλεόρασης κατά πόσο είναι αντικειμενικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ε, για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων είναι ένα ζητούμενο, αλλά η σημερινή κοινωνία αποδεικνύει ότι πολλές φορές τα εμπορικά μέσα προσδιορίζουν τις συνήθειες της νεολαίας και της κοινωνίας, οπότε και το περιεχόμενο της δημόσιας τηλεόρασης επηρεάζεται έμεσα και δεν είναι μέσα σε μία θερμοκοιτίδα στη σημερινή κοινωνία. Και το δεύτερο, η προσαρμογή της ε, τηλεόρασης στη νέα τεχνολογία, ψηφιακή κτλ. Είναι ένα ζητούμενο το ποιος θα κάνει και ποιος θα βοηθήσει τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση της προσαρμογής της δημόσιας τηλεόρασης, εάν αυτό αποτελεί κρατική ενίσχυση, εγκεκριμένη, αν είναι μέσα στο πακέτο, διότι η προσαρμογή των ιδιωτικών καναλιών μπορεί να γίνει με αύξηση του μερίσματος, διαμέσου των διαφημίσεων, διαμέσου των κερδών ενώ όταν κοπούν οι διαφημίσεις και κάποιες άλλες εισρωές θα πρέπει να δούμε πώς αυτές οι εθνικές ενισχύσεις είναι επιλέξιμες για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία που κοστίζει πολύ για τα μέσα τα κρατικά. Αυτά για ορισμένους προβληματισμούς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να περάσω τώρα στον ιδιωτικό τομέα, να φύγουμε από το δημόσιο, να πάμε στους, ε, στον κύριο Ross Bingham, Director, General Director of the Association of Commercial Television in Europe. Κύριε Bingham, για 10 λεπτά και ως ιδιωτικός τομέας που σέβεστε το χρήμα και το χρόνο, είσαστε just in 10 minutes. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παραστώ σήμερα στη συνεδρία σας. Μιλώ εκ μέρους των εταιριών που βλέπετε το σήμα τους αυτή τη διαφάνεια, VACT, ACT. Να πω ευθύ εξ αρχής ότι δεν μπορώ και δεν θέλω να μιλήσω για τον εμπορικό ραδιοφωνικό τομέα, ούτε για τον τύπο. Υπάρχουν και άλλοι που δεν τους εκπροσωπώ και θα πρέπει αυτοί να εκφραστούν σε αυτή τη συζήτηση ξεχωριστά από ποια έποψη μπορούμε να σχολιάσουμε εμείς το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης. Η σχέση που έχουμε εμείς, ιδιωτικός φορέας με τον δημόσιο τομέα. Από πού ξεκινάμε. Παρά τις επικρίσεις που ακούμε από πανεπιστημιακούς και άλλους. Ότι δημιουργείται δημόσια αξία και από το δημο... ιδιωτικό τομέα στην τηλεόραση. Παραδείγματα. Σε εθνικό περιεχόμενο προγραμματισμού είμαστε πρώτοι επενδυτές Υπάρχει μεγάλη συνεισφορά στον πλουραλισμό των μέσων από τα πολυ... την πολυκάναλη τηλεόραση και κάτι που ενδιαφέρει σαν πολιτικού ιδιαίτερο είναι ο ιδιωτικό τομέα που πρώτος είχε ειδησιογραφικά κανάλια 24 ώρε 24 ώρο, κυρίως στη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Τουρκία και την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε και στην Πορτογαλία. Αυτό είναι το ιστορικό. εμείς οι εμπορικοί φορείς πώ μπορούμε να, πώς μπορούμε να συνεπάρξουμε με το δημόσιο τομέα Sorry. Uh, right, uh, okay. I'm uh, maybe 11 minutes if I Ίσως 11 λεπτά αν πάω πιο σιγά, λέει ο κ. Μπικάνο. Λοιπόν, ε, δημιουργήθηκαν προσδοκίε, υπάρχουν προσδοκίε. Η συνύπαρξη λοιπόν μεταξύ δημοσίου τομέα και ιδιωτικού τομέα πάντα θα είναι κάτι δύσκολο. Δύσκολη σχέση. Υπάρχει τεράστιο δομικό όφελο σε ένα διτό, διπλό σύστημα. Αν η μία πλευρά παίρνει πάντα δημόσια χρήματα σε πολιετή βάση. Ε, μιλώ για χρήμα και ίσως μειώνω κάπως το επίπεδο, αλλά το καλό πρόγραμμα κοστίζει. Και, και στηρίζεται περισσότερο δημόσιο τομέα όσον αφορά του πόρους Αυτά είναι στοιχεία του 2006. Τι κάναμε στη διαφάνεια, σύγκριση κάνουμε στη διαφάνεια. Δημόσιου πόρου σε σύγκριση με τους ελεύθερους ε, σταθμούς του ιδιωτικού τομέα. Αυτά είναι στοιχεία του 2006. Τα στοιχεία του 2009 θα είναι ακόμα χειρότερα, πολύ χειρότερα για μας. Παράδειγμα, στη Γερμανία η δημόσια χρηματοδότηση ξεφερνά φέτος τα 8 δισεκατομμύρια στο δυτικό τομέα στη Γερμανία. Οι διαφημίσεις μειώθηκαν κατά 5% τον μήνα και 5% μείωση είναι καλή επίδοση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Um, Δεν ζητώ τη συμπάθειά σας ή δεν ζητώ ειδική βοήθεια ή θα φυλάξει κρατική επιχορήγηση για να μας στηρίξουν. Αλλά πιστεύω ότι με βάση αυτό το, την οικονομικό υπόβαθρο οι δημόσιοι, οι δημόσιοι πάροχοι δεν μπορούν να πούν αυτό που έλεγαν στο 8 Ιανουαρίου ότι τελικά ε, θα επικρατήσει ο ιδιωτικό τομέα και θα μονοπολίσει τα μέσα ενημέρωση. Αυτό δεν βοηθάει τη συνύπαρξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πάω σε πιο αισιόδοξη νότα. Υπό ποιε συνθήκε θα είναι πιο ορθολογική η βάση για τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο τομέων. Πρώτο στοιχείο. Συμφωνία όσον αφορά του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Ενώση και των κρατών μελών σχετικά με τον τομέα. Το θέμα ίσω να εξετάζεται περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε χρονικά. Όλοι θα συμφωνείτε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τον ρόλο να καθορίζουν ποια είναι η εντολή, τι καλύπτει ο δημόσιο τομέα όσον αφορά τι εκπομπέ. Κανεί δεν τα αφισβητεί, ούτε κι εμεί. Και επίση δεν συζητείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω αυτέ τι συνθήκε, εξασφαλίζει ότι και οι κανόνε περικρατικών επιχορηγήσεων και ενισχύσεων θα γίνονται σεβαστέ. Θα γίνουν σεβαστοί. Τι ζητάμε από τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να υπάρχει διακριτός προγραμματισμός που θα ελέγχεται από εξωτερική ρυθμιστική αρχή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ένα οικονομικό σύστημα που λειτουργεί. Η διπλή χρηματοδότηση, όταν παίρνουν ταυτόχρονα κάποιοι πάροχοι και ε, δημόσιες παροχές και έσοδα από τη διαφήμιση, είναι ό,τι χειρότερο, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους θεατές και για την κρατική τηλεόραση όταν υπάρχει ο συνδυασμός αυτός. Χώρες όπως η Γαλλία, η Τσεχία απομακρύθηκαν από τη διπλή χρηματοδότηση, δηλαδή διαφημίσεις και κρατική επιχορήγηση. Αλλά δημόσια χρήματα είναι καλύτερα για τη δημόσια τηλεόραση, διαφημίσει για την ιδιωτική τηλεόραση. Και η Γενική Διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής κινείται προ την κατεύθυνση. Κρατικέ επιχορηγήσει λοιπόν. Τώρα περνάμε για κρίση μάλιστα θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνε σχετικά με τι κρατικέ ενισχύσει και πρέπει να γίνεται σεβαστή επικουρικότητα. Αν εξετάσουμε το κείμενο τη κυρία Κρού, αν το διαβάσει κανεί προσεκτικά, εκεί αναφέρεται αρκετά επικουρικότητα. Δεν θα αναφερθώ σε όλε τι αναφορέ. 40 αναφορέ τουλάχιστον στι 106 παραγράφου αναφέρονται τόσες φορές η επικουρικότητα. Η, κρατική τηλεόραση. Ε, οι κρατικέ τηλεόρασει που είναι αντίθετες προς την κυρία Κρούς λόγω επικουρικότητας προστατεύουν εθνικά προνόμια είναι κατά του να ελέγχει η Κομισιόν μέσω τη Γενικής Διευθύνσεω της Αρμόδιας το πώς κινούνται. Ο έλεγχος εκ των προτέρων είναι η επικουρικότητα σε εφαρμογή σύσταση της Γενικής Διευθύνσεως Περιανταγωνισμού που αν την ακολουθεί τα κράτη-μέλη, τι σημαίνει, δεν θα παρεμβαίνει στη δημόσια τηλεόραση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, θα υπάρχουν προσφυγέ στον ιδιωτικό τομέα περί ανταγωνισμού αν υιοθετηθεί το κείμενο τη κυρία Κρού. Αν δεν υιοθετηθεί, θα υπάρχουν περισσότερε υποθέσει στα δικαστήρια περί ανταγωνισμού. Δεύτερη πρότασή μα για καλύτερη σχέση. Στάση συνεργασία και όχι μονοπωλίου από τη δημόσια τηλεόραση. Για να είμαι δίκαιος, στη Φλάνδρα στις 8 Ιανουαρίου βρέθηκε κάποια λύση. Δέχτηκαν τα ωφέλη της δημόσιας τηλεόρασης που συνεπάγεται ευθύνε όμως. Πρέπει να προσέχει κανείς τα συμφέροντα αλλωνών και να συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η συνεπαγωγή της κρατικής χορηγήσεως. Άλλες τηλεοράσεις κρατικές παραμένουν στον τομέα του μονοπωλίου. πρέπει να αλλάξει στάση. Όπως ας πούμε στα αθλητικά γεγονότα υπάρχει. Μπορεί να καλυφθεί από την κρατική τηλεόραση. Αυτό δεν το αφισβητούμε. Αλλά δεν μπορεί η δημόσια τηλεόραση να χρησιμοποιεί τα χρήματα του φορολογωμένου και να αγοράζει όλα τα δικαιώματα για τις αθλητικές εκδηλώσει και να μην μένει τίποτα για ιδιωτικό τομέα. Άλλη πρόταση. Να μιλούμε για διαφανή και αμερόληπτα στοιχεία και όχι για επιχειρήματα. στοιχεία, όχι επιχειρήματα. Κυρία Πρόεδρε, αναφέρθηκα σε θέματα που αφορούν περισσότερο την Οικονομική Επιτροπή. Θα καταλήξω σε κάνα δύο σημεία που αφορούν περισσότερο την Επιτροπή Πολιτισμού. Κυρίω η υποστήριξη του ευρωπαϊκού περιεχομένου. Αυτή η Επιτροπή τακτικά ακούει την κυρία Ρέντιν και διαπραγματεύεστε με το Συμβούλιο Υπουργών. Προσπαθείτε να πάρετε και το ελάχιστο ευρώ από τον υπολογισμό για να υποστηρίξετε τα μέσα ενημέρωση. Το υποστηρίζω αυτό θέλετε να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά χρήματα για δημόσιο ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Πολλά από τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιεί η κρατική τηλεόραση για να αγοράζει όμω σειρέ και ταινίε από το Hollywood. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Όμω κάποια κρατική τηλεόραση δημόσιευσε στοιχεία και είπε ότι 84% των χρημάτων για αγορά ταινιών χρησιμοποιήθηκε για αγορά αμερικανικών ταινιών από 70 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Εγώ εκτιμώ ότι για κάθε ευρώ που πάει για ευρωπαϊκά προγράμματα, 5, 6, 7 ευρώ πάνε προς Αμερική. Έχουν δικαίωμα ναι, να δείχνουν ταινίε οι κρατικέ τηλεοράσει, αόριστα, αλλά δεν πρέπει να στρέφονται όλα προ Αμερική. Λοιπόν, εσά Επιτροπή πολιτισμού και λέτε ότι μπορεί να υποστηριχθεί μέχρι το BMS ε, ο στόχος σας. Δεν θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ανεξάρτητα από το αν θεωρούμε ότι είναι λογικό εργαλείο, υπάρχει. Είναι κεκτημένο. Και πρέπει να συμμορφωθούμε. Και τα μέλη της ACT ε, είχαμε τουλάχιστον 66% ευρωπαϊκό περιεχόμενο και θεωρούμε γι' αυτό παράδεκτο ότι τρεις κρατικέ τηλεοράσει δεν συμμορφώθηκαν με την ποσόστοση όταν έγινε ο έλεγχος πρόσφατα. Κλείνω. Μη θέλοντα να συζητήσουμε TVWF, ε, αν μιλάμε πάντα αφηρημένα εμεί σαν τομέα, ε, δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας, δεν εξυπηρετούμε το στόχο μα. Οι κρατικέ τηλεοράσει αναφέρονται στην ποιότητα ε, του προγράμματος για, για πρόγραμμα που εντάσσει και συμπεριλαμβάνει με ευρύτερο κοινό. Καλό είναι αυτό, τα δημόσια χρήματα να δίνονται για αυτό το σκοπό. Πού διαφωνούμε στην πρακτική. Καθημερινά τι βλέπουμε. Ότι ο προγραμματισμός που συζητούμε, τα διακριτά προγράμματα, είναι περιθωριακά στο ωράριο, ίσως μετά τα μεσάνυχτα ή σε περιθωριακό κανάλι και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τα 22-23 δις κρατικής ενισχύσεως πηγαίνουν σε περιεχόμενο που δεν έχει αξία για το κοινό. Στην ACT το συζητήσαμε διεξοδικά, επί σειρά ετών, με την κρατική τηλεόραση. Το κάνουμε σήμερα, το ξανακάνουμε σε κάνα δύο χρόνια. Δεν πάμε πουθενά έτσι όμως. Διότι υπάρχουν πολλές ώρες προγραμματισμού στην Ευρώπη. Μπορεί να βρει παραδείγματα για κακά παραδείγματα κρατική τηλεοράσεω, καλά παραδείγματα κρατική τηλεοράσεω. Δεν βγαίνει άκρη. Οι μόνοι μπορούν να τα αναλύσουν σωστά, πώ χρησιμοποιούνται τα χρήματα του φορολογωμένου, είναι οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ μαζί με διάφορα αρμόδια δικαστήρια και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ανακοίνωση είναι σωστή δημιουργεί τη βάση για καλύτερη σχέση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ κύριε Μπίγκαμ. Ε, ευχαριστώ για, την, ε, για τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε ε, σχετικά για τη χρηματοδότηση της δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι, <clears throat> αν μπορώ να πω ότι αθέμητος ανταγωνισμός ε, στο θέμα τουλάχιστον των, ε, των οπτικοακουστικών με την κλασική οικονομική έννοια δεν υπάρχει. Διότι παρά τις ενισχύσεις τις οποίες έχει η κρατική τηλεόραση, βλέπουμε ότι το κοινό παρακολουθεί περισσότερο τα ιδιωτικά κανάλια, έχει μεγαλύτερη ακροαματικότητα από ότι η δημόσια τηλεόραση. Συνεπώς, ο ανταγωνισμός βρίσκεται επί του περιεχομένου και όχι τόσο για τη χρηματοδότηση. Και αυτό θέλω να το τονίσω γιατί εμάς εδώ μας ενδιαφέρει, όπως σωστά είπατε, το θέμα του περιεχομένου. Παρά τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις που γίνονται, το μειονέκτημα σε εισαγωγικά της κρατικής τηλεόρασης είναι ότι παρά τη χρηματοδότηση δεν έχει αντίστοιχη ακροματικότητα με βάση τα προγράμματα τα οποία καταθέτει. Και τονίζω ότι μία κρατική τηλεόραση στο περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι geographical ε, ή να δείχνει ζώα και ελέφαντες, αλλά να είναι και μία τηλεόραση με τέτοιο ποιοτικό περιεχόμενο που είναι attractive για τη σημερινή κοινωνία. Αυτό λοιπόν ε, για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα. Σχετικά με τα δικαιώματα για τον αθλητισμό, που είναι μία μεγάλη challenge για την κρατική τηλεόραση, θέλω να επισημάνω ότι το κόστος της αξίας των δικαιωμάτων για τα αθλητικά γεγονότα πλασματικά έχει ανέβει από τις ιδιωτικές τηλεοράσεις αγοράζοντας ή διαπραγματευόμενοι με τους φορείς, τους αθλητικούς φορείς, την αξία των δικαιωμάτων. Προφανώς αυτόν τον ανταγωνισμό μπαίνει και η κρατική τηλεόραση, αλλά το πώς διαμορφώνεται η αξία των δικαιωμάτων, ιδιαίτερα για τα αθλητικά γεγονότα, τα μεγάλα, Ολυμπιακούς, μεγάλα, τα ξέρετε εσείς οι άντρες, τα, τα sport events, ε, διαμορφώνουν μια πλασματική εικόνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και να περάσουμε τώρα στη, ε, ε, στη συζήτηση. Ανοίγουμε με την κυρία Χένικοτ και ακολουθεί η κυρία Ιερώνημη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες και μετά από αυτά που είπατε μήπως θα έπρεπε να θεωρήσουμε πέρα από, τις, από τα ποσοστά του τι συμπεριλαμβάνεται στην ιδιωτικό τομέα, τι στο δημόσιο τομέα, να κάνουμε και ανάλυση τι χρειάζονται οι ακροατές, οι θεατές. Καμιά φορά ο θεατής χρειάζεται μια παιδαγώγηση. Εάν βασιστούμε στην κρατική τηλεόραση για την ποιότητα, χρειαζόμαστε ιδιωτικά κανάλια που επίσης θα παράγουν ποιότητα. Διότι ο θεατής πριν βρει το σταθμό δεν θα πει «να ιδιωτικό κανάλι ποιοτικό, κρατικό κανάλι ποιοτικό, θα, το προϊόν που του προσφέρεται εξετάζει πρώτα. Δεν εξετάζει το που παρουσιάζει ο ιδιωτικό τομέα ή ο κρατικό. Οι θεατές χρειάζονται ποιότητα λοιπόν. Παιδαγωγική προσέγγιση, ισότητα, ισότιμη εκπομπή στην Ευρώπη, να βλέπει τι κυκλοφορεί στην Ευρώπη και να μπορεί να δει τι του προσφέρεται. Είναι πρέπει να υπάρχει και πληροφόρηση σωστή μέσω της τηλεόρασης. Οι τα κρατικά κανάλια έχουν ένα καθήκον δημόσιων υπηρεσιών. Έχουν ένα καθήκον αρχιοθέτησης και πάνω απ' όλα ε, έχουν την υποχρέωση της ανεξαρτησίας και την ε, αμερόληπτης ενημέρωσης και πλήρους και από αυτή την άποψη νομίζω ότι πολλά θα πρέπει να υποθούν. Διότι πολύ συχνά τα κρατικά κανάλια, τα ιδιωτικά κανάλια έχουν την επιτυχία που έχουν διότι η ενημέρωσή τους ίσως είναι διαφορετική. Δεν αρκεί λοιπόν απλώς να επιδοτείτε το κρατικό κανάλι για να προστατεύετε από κάθε κίνδυνο χρειάζεται να υπάρχει καλή ενημέρωση όσον αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση. Γιατί δεν σκεφτήκαμε το θέμα της επένδυσης, επένδυσης στο προϊόν. Αναφέρθηκαν οι πόροι που κατευθύνονται προς τα μίδια και τις ταινίες και τα μικρά προϊόντα πολιτιστικού περιεχομένου είναι δυσέβρετα για να προβληθούν είτε από ιδιωτικό ή δημόσιο κανάλι. Δεν βλέπουμε παραγωγούς προϊόντα ποιοτικά που θα περιέχουν προϊόντα κουλτούρας, ευρωπαϊκής κουλτούρας. Αν θέλουμε να περάσει ένα μήνυμα, εγώ έρχομαι από το διάλογο διαπολιτισμικού ε, ερχόμαστε από το έτος διαπολιτισμικού διαλόγου. Αν θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα διασυνοριακού διαλόγου, χρειάζονται προϊόντα οπτικοακουστικά για το ευρύ κοινό, ποιοτικά έργα, τα οποία θα μπορέσουν να διατεθούν μέσω των ιδιωτικών καναλιών και θα απευθύνονται βεβαίως και προς τα κρατικά κανάλια. Euh, λοιπόν, για τους ελέγχους είναι δύσκολο διότι αν Ευρώπη έχει κάποια κουβέντα να πει και αν θα πρέπει να το εθνική νομοθεσία η τηλεόραση ή θα πρέπει να εμπίπτει στην αρμοδία των κρατών μελών, αν πρέπει να συνεχιστεί αυτό, θα πρέπει να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την Ευρώπη για να υπάρχει και μια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το ερώτημα, τα κρατικά εθνικά κανάλια και τα ιδιωτικά κανάλια τα εθνικά, τι κάνουν για να στείλουν το ευρωπαϊκό μήνυμα να προβάλλουν την Ευρώπη. Εγώ δεν λέω πουθενά τέτοια προσπάθεια. Βλέπω γερμανική, ε, τις, τα, γαλλικά, τα γερμανικά νέα στην CDF, τα γαλλικά, γαλλικές ειδήσει στα γαλλικά κανάλια. Βλέπω το BBC που δίνει πληροφορίες ε, πολύ σύντομες, έχει ενημερωτικά δελτία σύντομα για να έχω πλήρη ενημέρωση για όλη την Ευρώπη είναι το Euronews που δεν το βλέπεις παντού. Μου μένει το Άρτε για τα γαλλογερμανικά. Διαφορετικά ε, παραμένω πεινασμένη. Ε, εκεί θα πρέπει συζητήσω το θέμα κατά πόσο μπορεί να κάνει κάτι η Ευρώπη να αλλάξει αυτή την κατάσταση και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία ε, Ιερώνημη, ε, Ρουθ, ε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τη θέση μου ως πρόεδρος και την ευκαιρία που έχουμε με τους, να ακούσουμε όλους τους προσκεκλημένους και θα ήθελα να αλλάξω λίγο την ημερήσια, τον τρόπο του, ε, της ακρόασης αν μπορέσουμε να ακούσουμε τους άλλους τρεις εμπειρογνώμονες προσκεκλημένους, γιατί νομίζω ότι τα ερωτήματα και τοποθετήσεις θα είναι συνολικές για όλους τους προσκεκλημένους και είναι και θέμα δικιάς μας φιλοξενίας εκ μέρους τους και να έχετε κι εσείς περισσότερο χρόνο να τοποθετηθείτε συνολικά στα ερωτήματα. Ε, εάν θα ήθελα λοιπόν να, με τη δική σας ε, βοήθεια θα ήθελα να περάσω στην, να δώσω το λόγο στην Μαρία Ρόν, Director Legal and Public Affairs, Danish Broadcasting Corporation. Ο χρόνος τυπικά είναι το 10 λεπτά για όλους. 10 minutes even for you. Thank you very much ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή που προσεκάλεσε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω μερικά πράγματα σχετικά με τον δικό μου κρατικό σταθμό. Ο DR δημιουργήθηκε το 1925 και είναι σχεδόν 100% χρηματοδοτούμενος από άδεια καταβολή εισφοράς για άδεια. Έχουμε το, το κρατικό κομμάτι είναι 70% και θα έχουμε περίπου 30% έχουμε στο σελίδα που καλύπτει πάνω 4% και έχουμε DAB, δηλαδή ψηφιακό ραδιόφωνο, δικτυακό ραδιόφωνο. Το TV2 δημιουργήθηκε το 1988 στη Δανία έχει πέντε κανάλια και μερίδι περίπου 40% καλύπτει. Το TV2 ήταν ε, χρηματοδοτήτο και μέσω αδείας που πλήρωναν οι θεατές και μέσω διαφημίσεων. Σήμερα μόνο μέσω συνδρομής και μέσω διαφημίσεων. Μετά την απόφαση για το TV2 πρέπει ακόμα να εξεταστεί ο ορισμός της κρατικής τηλεόρασης και πώς έχει αρμοδιότητα να ορίσει το πλαίσιο αυτό. Αν δει τη νομική βάση, είναι πολύ στερεή βάση. Επί σειρά ετών. Από τη συνθήκη ΕΟΚ, εδώ και 50 χρόνια ξεκίνησε, μετά έχουμε το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ πριν από 10 χρόνια και καταλήγουμε με την απόφαση για την TV2 μόλις πέρσι τον Οκτώβριο. Αυτή η απόφαση είναι σημαντικότατη διότι είναι η πρώτη φορά που το πρωτοδικείο ερμηνεύει τη νομική βάση περιορισμού της ε, κρατικής τηλεόρασης και των σχετικών υπηρεσιών που παρέχει. Τώρα, ποιος είναι ο ορισμός που περιέχεται στη νομική βάση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η εντολή της κρατικής τηλεόρασης είναι να εκπληρώνει δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες κάθε κοινωνίας και η διατήρηση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωση. Και πρέπει να είναι ανεξάρτητο το περιεχόμενο, να είναι ανεξάρτητης ο τρόπος ε, έκδοσης και ελέγχου του περιεχομένου. Και στην απόφαση TV2 ε, έγινε ξεκάθαρο ότι ο ορισμός κρατικής τηλεόρασης δεν συνδέεται με κάποια πλατφόρμα τεχνολογικής τεχνολογική πλατφόρμα εκπομπής, αλλά βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα να καθορίσουν τι ακριβώς κάνει αυτή η κρατική τηλεόραση, ποιο είναι το, η εντολή που τους δίνεται. Για μας είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η απόφαση χρησιμοποιεί λέει ότι τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα να καθορίσουν ποιοτικά, γενικά και από πλευρά ποιοτική τι είναι η κρατική τηλεόραση. Τι άλλο υπογραμμίζει η απόφαση. Ότι η μέθοδος χρηματοδότησης δεν έχει σχέση με τον ορισμό και ακόμα πιο σημαντικό της, εμπορ... της κρατικής τηλεόρασης και οι δραστηριότητες των εμπορικών φορέων δεν παίζουν ρόλο για τον καθορισμό της εντολής. Και μπορεί να ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον καθορισμό που κάνει το κράτος μόνο για σφάλματα. Στην νομοθεσία της Δανίας η εντολή του TV2 ε, είναι αυτός που φαίνεται στη διαφάνεια. Μέσω τηλεοράσεως, αδιοφώνου, διαδικτύου κλπ. Το TV2 Πρέπει να παρέχει ευρύ φάσμα προγραμμάτων και υπηρεσιών, να δίνει ειδήσει, ε, γενική ενημέρωση, ψυχαγωγία, χρειάζεται επικοινομορφία και ποιότητα στον προγραμματισμό. Στην απόφαση για την TV2 είναι ξεκάθαρο ότι είναι συγκεκριμένη η εντολή που δίνεται και ανταποκρίνεται στη νομική βάση. Τώρα, αν δείτε το σχέδιο ανακοινώσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπετε ότι εδώ εισάγεται λεπτομερής διαδικασία για να καθορίσει την εντολή του κρατικού καναλιού. Ε, επεκτείνονται οι φυστάμενες δραστηριότητε, αλλά εισάγονται και νέες υπηρεσίες. Για μας είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό δεν αντιστοιχεί στην απόφαση για το TV2, για το TV2 και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ασχολούνται με το θέμα, να καθορίζουν δηλαδή ποιε είναι οι δημόσιε υπηρεσίε που παρέχονται από την κρατική τηλεόραση. Και είναι σαφέ για μα ότι αυτά που εισάγονται στο σχέδιο ανακοίνωση, δηλαδή η μέθοδο χρηματοδοτήσεω ή πόσα αμείβεται το προσωπικό ε, και τα σχετικά κριτήρια δεν αντιστοιχούν στην απόφαση TV2. Και το πιο σημαντικό ίσως σχετικά με αυτό που συζητούμε σήμερα είναι το τρίτο κομμάτι, εκεί στο κάτω μες διαφάνειας, ότι το σχέδιο ανακοινώσεως εισάγει εκ των προτέρων αξιολόγηση. Δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση συνεπιών για την αγορά, για, την κρατική, για τον κρατικό πάροχο και σχετικά κριτήρια. Αν γίνονται δημόσιες εάν είναι δημόσια προσφορά των υπηρεσιών ή υπάρχει ενδεχόμενο εμπορική εκμετάλλευση αυτών. Αυτό δεν αντιστοιχεί στην απόφαση TV2. Και επίση, αναφέρεται σαφώ ότι αν εισαχθεί αυτό το μέτρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι στερεί κανεί τα κράτη-μέλη από την εξουσία να καθορίζουν τι αποτελεί δημόσια υπηρεσία. Δημόσια παροχή υπηρεσιών μάλλον. Το συμπέρασμα για μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να περιορίσει τα κράτη-μέλη, τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να καθορίσουν την εντολή τη παροχή δημοσίων υπηρεσιών μέσω εισαγωγή νέων στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα των εμπορικών φορέων. Και επίση δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει λεπτομερείς ε, υποχρεώσεις για τον καθορισμό όλων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε το εξής η αρχή της επικουρικότητας και η εθνική ποικιλομορφία πρέπει να γίνουν σεβαστά. Ταυτόχρονα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά ρυθμίσεως. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντική η ρύθμιση όταν εισπράττει κανεί ένα τέλος από την άδεια, από τη συνδρομή και ότι έχει ένα δημόσιο καθήκον που πρέπει να εκπληρώσει. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό κυρίως για τις μικρές χώρες είναι ο εθνικός νομοθέτης να, να αποφασίζει και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς της χώρας και τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας. και σχετικά με αυτό πρέπει να πω ότι στη Δανία έχουμε ήδη μία δοκιμή για τις δημόσιες αυτές αξίες από αρχές Ιανουαρίου 2007. Αλλά λαμβάνει υπόψη ότι είμαστε μικρή χώρα και ότι μικρή γλώσσα και μικρή αγορά συνολικά. Είναι πολύ σημαντικό για την κρατική τηλεόραση, για τους κρατικούς παρόχους, η εντολή να μην καθορίζεται σε σχέση με την αγορά. Και είναι σημαντικότατο επίσης να καθορίζεται αυτό με έναν τρόπο τεχνολογικά ουδέτερο, ούτως ώστε ο δημόσιος πάροχος να μπορεί να αναπτύσσει τις δικές του διασυνδέσεις με την τεχνολογία. και να ακολουθεί και το κοινό που πολλές φορές μπορεί να προχωρά τεχνολογικά. Οι θετικές συνέπειες θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι θετικές συνέπειες της κρατικής τηλεόρασης των κρατικών παρόχων. Θα πρέπει να ανέβει ο πύχης για την ποιότητα των προγραμμάτων που παρέχουν οι κρατικές τηλεοράσεις. Συχνά χρησιμοποιούμε νέα τεχνολογία και ξεκινάμε, είμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την νέα τεχνολογία και υποστηρίζουμε καλλιτεχνικό περιβάλλον, ποιοτικό περιβάλλον, το οποίο βέβαια ωφελεί και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. <clears throat> Ήταν πραγματικά μια άλλη διάσταση για το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης και για τον τρόπο χρηματοδότησης, ε, για το ρόλο του κράτους ε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν προσπαθεί να ορίσει ορισμένα κοινά κριτήρια κρατικών ενισχύσεων και φυσικά παραμένει πάντα ανοιχτό και περιμένουμε και μία απάντηση στα πλαίσια της συζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο μια δημόσια τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιεί τα αποθεματικά τα οποία υπάρχουν από τα δικαιώματα, ένα, αλλά και τον τρόπο διαφάνειας των κρατικών ενισχύσεων, διότι, εν πάση περιπτώσει, το θέμα της διαφάνειας είναι το α και το ω σε μια υγιή οικονομία. Ε, θα ήθελα να περάσω στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Αλεξάνδερ ε, Βράμπετς, ε, Director General of ORF, για 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Εξωτερικέ κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σα. Να σα αποτείνω εδώ το λόγο. Η ORF είναι η εθνική ε, ε κανάλια της ε, ε, Αυστρίας τηλεόραση, ραδιοφωνία και μία υπηρεσία online. Είμαστε ηγέτε στην αγορά σε όλου του τομεί. Έχουμε όμω μια ειδική κατάσταση στην Αυστρία, ιδίω όσον αφορά την τηλεόραση, ότι είμαστε μια μικρή χώρα, 8 εκατομμύρια κάτοικοι, που μέσω τη αριθμοποίηση είμαστε τμήμα τη γερμανική αγορά ΜΜΕ. Το 95% των νοικοκυριών στην Αυστρία μπορούν να ε, δέχονται τα γερμανικά προγράμματα στην ίδια γλώσσα, α πούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ΟΕΡΕΦ και για τις ιδιωτικές ανταγωνιστικές εταιρείες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, γι' αυτό στη συζήτηση ε, λέμε ότι θα πρέπει να διακανονίζονται οι ε, δημόσιες υπηρεσίες από τον εθνικό νομοθέτη γιατί υπάρχουν ακριβώς τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις αγορές τη ραδιοφωνία και τηλεόραση στην Ευρώπη. Οι μικρές χώρες έχουν άλλες ανάγκες και άλλα προβλήματα ή, από ότι μεγάλες χώρες ή χώρες όπως απο οτι μεγαλες χωρες η χωρε οπω η αυστρια που είναι τμήμα ενό μεγαλύτερου γλωσσικού χώρου. Αυτά και μέσα στα πλαίσια της επικουρικότητα, τα οποία υποστηρίζω εδώ. Το δεύτερο, πάλι λόγω του ότι είμαστε μικρή αγορά, ε, παίζει σημαντικό ρόλο για την ε, κινηματογράφο στην Αυστρία. Το 90% των προγραμμάτων τα παράγει ο ΡΕΦ εν μέρη και σε συνεργασία με δημόσιους εκπομπέας της Γερμανίας. Δηλαδή χωρίς την ΟΕΡΕΦ δεν θα υπήρχε καθόλου μια ε, λειτουργούσα αγορά κινηματογράφου στην Αυστρία. Και εδώ έχουμε λοιπόν ειδική ευθύνη. Είναι σαφές και ελέγχθη πλειστάκης ότι ο ευρωπαϊκός δημόσιος, οι ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης ε, υποτελούν ένα πολιτισμικό αγαθό. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πρόγραμμα για μικρές ομάδες στόχου, αλλά ένα πρόγραμμα που να στρέφεται προς όλους τους πολίτες έχει σαν στόχο βέβαια την ενημέρωση και τον πολιτισμό που μπορεί να εκπληρώσει το έργο αυτό εάν ενταχθεί σε πιο ευρύ ε, πεδίο προσφοράς στον αθλητικό και στον ε, ψυχαγωγικό τομέα. Επίσης, χρειαζόμαστε γι' αυτό ευρεία προγράμματα ψυχαγωγικά γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να ε, δούμε να συμμετέχουν πολύ και να τους ενημερώσουμε και όλες κατάλληλα. Ε, στην Αυστρία σχεδόν όλα τα νοικοκυριά έχουν περάσει στο διαδίκτυο τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του ε, υπολογιστή και γι' αυτό θα πρέπει να αντιδράσουμε στην, στον κατακαιρματισμό της αγοράς, συμπληρώνοντας τα κύρια προγράμματα. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα και την υποχρεώση να στρεφόμαστε προς όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Θα πρέπει δηλαδή γι' αυτό να έχουμε τη δυνατότητα ιδίω να στραφούμε και να προσελκύσουμε και τους νέους. Πράγμα που σημαίνει ότι στις online πλατφόρμες που δημιουργούνται θα πρέπει να είμαστε ανάλογα παρόντες. Αυτό σημαίνει ότι τώρα μετατοπίζεται η διάσταση του αναγωνισμού. Τα τελευταία ε, δέκα χρόνια συζήτηση μεταξύ των δημοσίων ε, ε, εταιριών και του ECD ήταν πάρα πολύ έντονη. Τώρα όμως έχουμε νέους ανταγωνιστές από τον τομέα Brent ιδίως. Υπάρχουν εδώ πέρα επίσης κάποιες ε, διαφορές και με τον τομέα των εντύπων μέσων που υπόκεινται μεγάλες αλλαγές αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να δουν ότι δεν υπάρχει εδώ πραγματικός αναγωνισμός. Ο πραγματικός αναγωνισμός ε, στις νέες υπηρεσίες προέρχεται από τον τομέα των μη μη ε, νέες εταιρείες όπως η Google, Φερρυπίν, Facebook και άλλα ή από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών δηλαδή όχι από τον τομέα των ΜΜΕ και αυτό θα είναι μια πρόκληση σε όλα τα διακονιστικά βήματα να έχουμε κατά νου ότι στο διτό σύστημα δεν πρέπει να δημιουργήσουμε διακανονισμούς που να προασπίζουν τα δικαιώματα των εντύπων μέσων παραδείγματο χάρη ή του ανταγωνισμού μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών και που θα ωφελήσουν εκείνους που δεν υπάρχουν σε κανένα διακανονισμό και θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι το 90% των ταινιών που δείχνονται ε, προέρχονται από εκτός της Ευρώπης. Το ίδιο ισχύει και για αυτές τις εταιρείες στις οποίες αναφέρθηκα Google κλπ. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. time θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε ε, Μπράμπεκ, ε, και πραγματικά το θέμα το οποίο θίξατε ότι ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως διαμέσου των νέων τεχνολογιών οι οποίες προκύπτουν, το ψηφιακό μέρισμα, το online, είναι ένα καινούριο μοτίβο ανταγωνισμού το οποίο ισότιμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει και η δημόσια τηλεόραση και η ιδιωτική ε, και να μην περιοριστούμε απλά και μόνο σε παραδοσιακές μορφές οικονομικού ανταγωνισμού. Ε, θα ήθελα να δώσω τώρα στον ε, τελευταίο προσκεκλημένο μας, στον κύριο Πασκάλ Άλμπερτ Κύρχιντα, ε, πιθανά να χρειάζεται υπότιτλους για Ελληνίδα να βάλω για να πω το όνομα, πιστεύω να, να το είπα αρκετά σωστά, είναι Head of the ZDF, Europe Office Brussels και σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γερμανικά, αλλά οι διαφάνειές μου είναι στα αγγλικά. Ναι, λέγομαι Πασκάλα Απρικέχινερ, εκπροσωπώ του CDF, του δεύτερη μεγάλη υπηρεσία τηλεόραση στη Γερμανία. Και Επίτροπος, κύριε Ρέντινγκ, είπε πριν σε μια εβδομάδα σε μια συνέντευξη Πώς θα ήθελα να κοιτάει την τηλεόραση το 2020. Σίγουρα θα είμαι ο διευθυντής του δικού μου προγράμματος. Θα κοιτάω εκείνες τις εκπομπές που μου φαίνονται πιο ενδιαφέρουσες και όποτε εγώ το θέλω. Με αυτά η Επίτροπος πραγματικά είπε κατά λέξη αυτά που ενδιαφέρει τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από αυτήν σε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα του 2007 αναφερθήκανε στα μέσα δημοσίων υπηρεσιών την εποχή αυτή ότι η δηλητική τηλεόραση είναι περισσότερο από την κλασική τηλεόραση. Χαίρομαι που η Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να συζητήσουμε συζητήσουμε το θέμα της αναθεώρησης οδηγίας αυτής μέσα σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Η οδηγία αυτή για τα ΜΜΕ αποτέλεσε έναν ακρογωνιαίο λίθο για τον διαγωνισμό των ΜΜΕ στην Ευρώπη που θα πρέπει στο μέλλον να προσανατολίζεται στην, ε, στο περιεχόμενο τους και ανεξάρτητα από τον τρόπο διάδοσης. Η ανακοίνωση του 2001, στην οποία αναφέρομαι, είναι μια ανακοίνωση που μας ικανοποιεί ακόμα. Και γιατί. Γιατί προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζεται για να αντιδράσουμε στις ε, ε, εξελίξει της αγοράς και αφορά τρεις ε, πτυχές. Την εξελικτικό χαρακτήρα της ε, ραδιοτηλεόρασης, τον λειτουργικό χαρακτήρα της δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεόρασης και τρίτον την αυτονομία των κρατών μελών όταν ορίζουν την εντολή τους και όταν χρηματοδοτούν. Γιατί θα έπρεπε η ανακοίνωση αυτή να αναθεωρηθεί Δύο λόγια αναφέρανται Γιατί είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο, υποτίθεται. Καταρχήν τεχνολογική εξέλιξη και δεύτερον το γεγονός ότι υπάρχουν στρεβλώσεις της αγοράς από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτά είναι τα σημεία που θα ήθελα να εξετάσω μαζί σας και να δούμε κατά πόσον αυτή η ανησυχία είναι δικαιολογημένη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι υπερβολική η ανησυχία αυτή. όσον αφορά την στρέβλωση των αγορών όπως είπα στις υπηρεσίες ε, ραδιοτηλεόρασης και όσον αφορά την τεχνολογική εξέλιξη ε, όποιος το σκέφτεται αυτό δεν σκέφτεται λειτουργικά και σφαιρικά. Για να εξετάσουμε το παρελθόν. <laughs> Τι είναι η ραδιοφωνία. Αυτό είναι ραδιοφωνία του 1920. Επί δεκαετίες μόνο ραδιοφωνία υπήρχε όταν λέμε εκπομπές. 30-40 χρόνια αργότερα εκπομπές είναι οπτικές. Και μετά περνάμε στο έγχρωμο. τέλετεξ τη δεκαετία του 70. Ίντερνετ και κατευθυμία τηλεόραση εδώ και αυτή είναι η μορφή σήμερα. Θα πρέπει να ρωτηθούμε Τι είναι το καινούριο στη σημερινή εξέλιξη, γιατί αυτό που ήταν πάντα όσον αφορά τις εκπομπές ήταν ότι ήταν ε, συγκλητικό, ανεξάρτητο από την τεχνολογία κατά κάποιον τρόπο, ουδέτερο όσον αφορά την τεχνολογία και εξελικτικό συνεχώς. Αυτό που είναι σήμερα μεγάλη πρόκληση είναι η σύνδεξη, η τεχνολογική της πλατφόρμας και της διαδικασίας παραγωγής και το όφελος που μπορεί να έχει ο θεατής. Γιατί ο θεατής ε, βλέπει συγκλήσιμες υπηρεσίες. Αυτό βέβαια δυσκολεύει στην πραγματικότητα την διάκριση μεταξύ του παλιού και του νέου. Και μάλλον και τη διάκριση μεταξύ του γραμμικού και του γραμμικού. Μακροπρόθεσμα. Η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η ραδιοτηλεόραση σήμερα θα ήθελα να στην εξετάσταση μαζί σας. Κυρίως η τηλεόραση είναι το πιο διαδεδομένο ηλεκτρονικό μέσο, αλλά στην Γερμανία τουλάχιστον, από την τελευταία, ε, μετά την τελευταία ε, ποδοσφαιρική, ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, μειώνεται αυτό, προχωράει πολύ περισσότερο το διαδίκτυο. Ξέρουμε ότι τώρα πια 100% των 14-29 ετών, των νέων 14-29 χρησιμοποιούν το διαδίκαιο. Υπάρχουν όμως αδύνατες ομάδες, ε, συμπεριλαμβάνουν και εκείνο που είναι πέρα των 60. Και το 2008 στην γερμανική αγορά τουλάχιστον Ε, χρησιμοποίησαν ε, περισσότερο το διαδίκτυο από την τηλεόραση αυτή Αυτοί νέοι των 14-29 ετών. Παρόλο που το μεγαλύτερο ρόλο εξακολουθούν να παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα, βλέπετε ότι έχουμε και τα, τις πύλες ε, βίντεο και τα βίντεο γενικά, όσο πάει και περισσότερο ρόλο στη χρήση του διαδικτύου. Πράγμα που έχει επίδραση στην τρόπο χρησιμοποίησης από τους χρήστες. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει από την άλλη μεριά να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθούν υπόψη και να λάβουν υπόψη τις συνήθειες ε, παρακολούθησης. Δηλαδή εμείς είμαστε μια οικογένεια, όσο μόνο το κύριο κανάλι αλλά και άλλα κανάλια για να μπορούν όλοι να μας ε, βλέπουν όπου βρίσκονται και βέβαια και μια δικτύωση με τις υπηρεσίες online. Το κυριότερο που κάναμε εμείς ήταν η Mediatek για το λεγόμενο Ketchup TV. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλό, ε, υψηλή προσφορά ενημέρωσης και βλέπετε από την άλλη μεριά όσον αφορά τη χρήση ότι το εικονικό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από δική μας σκοπιά είναι καλά τα πράγματα. γιατί μπορούμε να τοποθετήσουμε στη ιδιαίτερη αυτή μόνο τη δική μας παραγωγή. Θα ήθελα να σας δώσω ένα ε, παράδειγμα όσον αφορά την cross-media χρησιμοποίηση όλων των μέσων δηλαδή. Πέρσι προ... είχαμε παράγει μια ε, δεκαμερή ε, παραγωγή, η Γερμανή λεγόταν, είχαμε 16% οραματικότητα θεαματικότητα, πάρα πολύ σημαντικό, 11,6 μεταξύ των νέων, 14-29 δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από τη συνήθως, συνήθως είμαστε στα 7. 9 εκατομμύρια σελίδων ετυπώθηκαν από το συνοδευτικό υλικό και 3 εκατομμύρια ketchups. Ε, guter ε, από ό,τι βλέπετε, ε, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού χρησιμοποιεί αυτό το cross-media. Μιλάμε δηλαδή για πραγματικότητα, όχι για όραμα προς το μέλλον. Δεύτερο σημείο. Κάθε φορά που δημόσιες υπηρεσίες καλύπτουν νέο τομείς υπάρχει πάντα μια καταγραφή. Εγώ δεν μπορώ παρά να σας αναφερθώ στην γερμανική αγορά για να δούμε την ψηφιακή αγορά στην ε, Γερμανία και την κλασική αγορά τηλεόρασης. Βλέπετε ότι η γερμανική αγορά είναι μια αγορά στην οποία δεν φτάνει κανείς το 20-25% είναι μια κατακαιρματισμένη αγορά πράγμα που είναι ενοχλητικό για την ιδιωτική μας, για τους ανταγωνισμούς μας αλλά βλέπετε ότι στην ψηφιακή αγορά αριστερά είναι, ε, δεξιά είναι αυτό, μειώνεται το ποσοστό, ενώ για την ΕΡΤΕΛ αυξάνεται. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά αριθμητικά στοιχεία. Ο Ρος ε, είχε μια διαφορετική εικόνα νομίζω. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι εγώ έχω αναφερθεί μόνο στα έσοδα από την τηλεόραση, όχι μόνο και αυτά του ε, ραδιοφώνου. Και έχω προσθέσει και την Pay TV που την είχε αφαιρέσει νομίζω ο Ρος προηγουμένως, γι' αυτό διαφέρουν οι εικόνες μας. Όσον αφορά τα τέλεια διαδόθησης, έχουμε μια αύξηση περίπου 1,46% ανά έτος. Πολύ λιγότερο από τα κέρδη των ιδιωτικών ανταγωνιστών μας, οι οποίοι έχουν 85-90% της αγοράς ε, διαφήμισης. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν δημοσιεύουν τα στοιχεία αυτά. Τα δικά μας ψηφιακά κανάλια και οι υπηρεσίες online δεν ε, ε, καλύπτονται από διαφημίσεις. Ξέρετε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα τους εμφάνισης online για τις ειδήσει. Έχουμε κάποια προβλήματα με τους εκδότες. Έχουμε εδώ ένα παράγουμε από τη Voda Media που το 2006 είχε 230 εκατομμύρια ευρώ στην ψυχική αγορά, πάνω από 14% της αγοράς του. Το ZF Online αυτή τη στιγμή έχει ένα ετήσιο προπολογισμό μεταξύ 2009-2012 12 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, χωρίς το κόστος μετα... αναμετάδοσης στην αγορά τηλεόρασης που είναι σημαντική για τους ε, ανταγωνιστές μας 14-29 ετών είπαμε είναι αυτοί οι άνθρωποι δεν φτάνουμε ούτε στα 25 και αυτό που είναι σημαντικό στην αγορά ενημέρωσης έχω εδώ κάποια αριθμικά στοιχεία το Heute.de είναι οι ειδήσει μας κάθε βράδυ. 5 εκατομμύρια επισκέψεις ε, υπάρχουν. Βρισκόμαστε 13η σειρά δηλαδή. Και άμα κοιτάξετε Spiegel Day και Bill βλέπετε ότι τα αριθμικά στοιχεία είναι πολύ πολύ πολύ ψηλότερα. Και άμα πάρει το σύλλογο της αγοράς αυτής έχουμε λιγότερο από 2% μερίδιο. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ να αναφερθεί κανένα σε ε, καταφανή στρέβλωση του αναγνωσμού. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιείται πάντα και στη Γερμανία ιδιαίτερα. Υπάρχει βέβαια και ο γενικό περιορισμός που έχουμε για τι νέε μας υπηρεσίε, δηλαδή περιορισμός ε, παραμονής για αυτό που προσφέρουμε, να υπάρχει μια, ένα σχετισμό με το πρόγραμμα, υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί που του ανέφερα και βέβαια και έχουμε και αυτό το τεστ τριών ε, βαθμίδων που αναφέρθηκε και προηγουμένω. Και εδώ μία σύντομη πρόταση του Ματία Ντόφνερ, του επικεφαλής ε, του εκδοτικού του οίκου Σπρίνγκερ, όσον αφορά τον ορισμό τη αγορά και τον αναγνωρισμό στο οποίο μιλάμε. Η κυρία Βασιλή το αναφέρθηκε, ανέφερε προηγουμένω, είπε σε μια συνέντευξη πέρσι ότι ίσω η ευέλεια, η ψηφιακή των δημοσίων υπηρεσιών είναι τεραμαράσια, αλλά δεν μπορεί να αντικαταπτουριστεί σε χρήμα διότι δεν έχουμε ακριβώ έσοδα από διαφήμιση. Λοιπόν, δεν θα μπορεί έτσι να βλαφτούν οι ιδιωτικοί ε, σταθμοί. Είναι σωστό ε, εδώ για τακτικούς λόγους ε, συγκρίνονται τα σύγκριτα. Μίλαμε μαχλάδια, όπως λέμε. Και αυτό για να αποκλειστούν προφυλακτικά οι ανταγωνιστές. Τελειώνω σιγά σιγά. Δεν τίθεται θέμα κυρίε και κύριοι ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ισχύουν και για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, αλλά η εφαρμογή του ανταγωνιστικού δικαίου αυτού πρέπει να εφαρμόζεται, να είναι μόνο εκεί που ε, ε υπάρχει κάποιος λόγος να εφαρμοστούν, όπου υπάρχει δηλαδή πραγματικά ανταγωνισμός και πιστεύουμε ότι το θέμα αρχής όσον αφορά και τα νέα μέσα και των διαγωνισμών θα πρέπει να είναι ποια είναι η ισχύ τους, η εμβέλειά τους, πόσο ενήμερα είναι, πόσο επίκαιρα είναι και εάν φτάσουμε σε νέα διατύπωση του κειμένου του 2001 θεωρούμε ότι όσον αφορά το προσχέδιο που ξέρουμε του Γενουαρίου του 2009 δεν θα μπορούμε κατά τον ίδιο τρόπο να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ παλαιού και νέου, γιατί αυτό ούτε είναι σύμφωνο με μια δοτερότητα τεχνολογία, ούτε με τι πραγματικέ εξελίξει που σα προανέφερα. Θα πρέπει λοιπόν ο εξελικτικό χαρακτήρας των συγκλίνων μέσων να ληφθεί υπόψη. Και το ίδιο ισχύει και για τον ανταγωνισμό των ε, ειδήσεων αυτό το κριτήριο θα πρέπει να ληφθεί πολύ πιο έντονα υπόψη και συμμερίζομαι απόλυτα αυτό που είπε και η Δανή συνάδελφο προηγουμένου για την TV2 στη Δανία και τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου. Τέλος, αλλά βέβαια πολύ σημαντικό, η μόνη ύπαρξη και δραστηριότητα των δημοσίων υπηρεσιών δεν αποτελεί αυτή καθ' μια στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε κατά τη γνώμη μου ότι αυτοί οι διακονισμοί που συζητάμε σήμερα θα πρέπει πάντα να εξεταστούν μέσα στο συνολικό πλαίσιο. Δηλαδή ποια είναι τελικά η εικόνα στην Ευρώπη για τα ΜΜΕ που θέλουμε να έχουμε. Και θα ήθελα να αναφέρω, να παραφέρω στο κάτι που είπε ο κύριος Μπούρντα, που τα Μπούρντα Μέτι εν Deutschland, που είπε πριν από μερικέ εβδομάδε ότι ενώ ο ανταγωνισμό μα προηγουμένω ήταν Γκρουνουριάρη, Σπίγελ, σήμερα είναι Google. Γιατί αν εμεί έχουμε χίλιες, επαφέ επαφές με τον καταναλωτή, το Google έχει ένα εκατομμύριο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Αυτό θα πρέπει να είναι το μέτρο με όλο το σεβασμό βέβαια προς τους κατά βάση κανόνες του δικαιών ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Πασκάλ, θέλω να σε ευχαριστήσω για την εισήγησή σου. Ε, δεν τολμώ να επαναλάβω και πάλι το επίθετο. Μου επιτρέπεις να λέω Πασκάλ. Ε, και πραγματικά νομίζω ότι <clears throat> ε, έθεσες ε, πραγματικά τη διάσταση του υγιούς ανταγωνισμού ε, με την ε, κρατική δημόσια τηλεόραση, του ρόλου, της νέας τεχνολογίας και νομίζω ότι η παρουσίαση του ZDF δίνει μία προπτική και στη συζήτηση την οποία έχουμε να καταθέσουμε εμείς σαν Επιτροπή Πολιτισμού αλλά και σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Ε, θα ήθελα τώρα να συνεχίσω τη ε, την ε, συμμετοχή των αγαπητών συναδέλφων. Ιερώνυμη, έχεις το λόγο. Καταρχήν έχω μια ερώτηση όσον αφορά τη διαδικασία. Για τη διαδικασία λέω έχω μια ερώτηση κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν βλέπω κανέναν εδώ από την Γενική Διευθυνσία Ανταγωνισμού δεν εκπροσωπείται. Εδώ όλοι το, τα έδρα της Κομισιόν δεν υπάρχει κανένας. Θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια της ε, διοργάνωσης αυτής της ημερίδος είχαμε καλέσει και την Επιτροπή και τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής. Η ημερίδα αυτή, η ακρόαση, είναι ανοιχτή για όλους τους συναδέλφους και για τα μέλη της ΕΚΟΝ, της Οικονομικής ε, Επιτροπής. Ε, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι θέμα συμμετοχής. Ο καθένας τι θέλει να ανοίξει. Sorry. Ruth. Dann äh, möchte ε, τότε θα ήθελα ξεκάθαρα να πω εισαγωγικά το εξή. Η Επίτροπη Ρένιγκ είπε ότι περιμένει η ανακοίνωση όπως το 2001 να προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και τη Γενική Διεύθυνση για την Κοινωνία της Πληροφόρησης. Από κοινού και αυτό συμφωνώ απόλυτα και το τονίζω και προς όφελος του διτού συστήματος ραδιοτηλεόρασης και το θεωρώ για αυτούς τους λόγους απαραίτητα. Τώρα, επί Είναι σαφές χρειαζόμαστε τις διευκρινήσεις της εντολής, τη διαφάνεια της χρηματοδότησης. Αυτά όμως είναι όλα θέματα που ήδη υπάρχουν στην ανακοίνωση του 2001. Νέο θέμα για την αιτιολόγηση της ε, πανεξέτασης ανέφερε η Κομισιόν τις νέες τεχνολογίες και τις επιπτώσεις από τη σύγκληση. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην ερώτησή μου σε αυτά και να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν προς την κυρία Ρορμπιρόν. Βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες και κυρίους για τις ε, πληροφορίες που μας δώσαν και τις ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις τους. Αλλά θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση συμπληρωματική, γιατί θεωρώ ότι για το Κοινοβούλιο και για την Κομισιόν βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιο είναι το σημερινό επίπεδο απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και γι' αυτό σας ρωτώ, μπορείτε να συμπεριλάβονται αυτές τις έννοιες, δηλαδή το κατά πόσο είναι σημαντικό για την αγορά, κατά πόσο είναι αποτύχανη η αγορά. Γιατί στην αρχική πρόταση της Κομισιόν είχε, υπήρχε και αυτή η αποτυχία της αγοράς. Εμείς είπαμε ότι ο έλεγχος θα πρέπει να είναι ο έλεγχος της κατάχρησης. Και βέβαια αυτό που είναι σημαντικό είναι και οι επιπτώσεις στην αγορά, το marketing impact. Ίσως αυτός ο όλυχος της κατάχρησης, επίπτωση της αγοράς και αποτυχία της αγοράς. Αυτά ίσως θα μπορέσετε να μας παρουσιάσετε. Να ξέρουμε ποια ήταν τα μηνύματα του δικαστηρίου σχετικά. Η δεύτερη μου ερώτηση θα ήθελα να την αποτείνω στον κύριο Ζαπιό που αναφέρθηκε στη δυτή εξέλιξη των ΜΜΕ. εν και των νέων ψηφιακών μη γραμμικών υπηρεσιών. Ελέγχθη προηγουμένως στα οδηγία για τα οπτικοστικά μέσα. Είπαμε ξεκάθαρα. Αποχωρήσαμε από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εσείς στη Γαλλία πώς εξηγείτε τις γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίες σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον αποχωρισμό από αυτά δηλαδή κάποιες υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο δίκαιο ραδιοτηλεόρασης. Λόγω στον κύριο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα. Παρόλο που είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σαφές όμως ότι για πολλά κράτη-μέλη και για το Κοινοβούλιο αυτό το θέμα, αυτό το σχέδιο ανακοινώσεω δεν μπορεί να θετηθεί του το τρόπος. Και λυπούμε ω μέλος της Οικονομικής Επιτροπής που η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό δεν είναι εδώ. Χαίρομαι το Συμβούλιο είναι εδώ. Χαίρομαι που αρκετά κράτη-μέλη εκπροσωπούνται εδώ. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικότατο μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα όσον αφορά το μέλλον των δημοσίων φορέων παροχή υπηρεσιών, χρειάζονται νέα τεχνολογία, είναι σαφέ και χρειάζονται επίσης και αλλαγή από γραμμικές σε μη γραμμικές υπηρεσίες. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο για να μπορούν οι δημόσιοι πάροχοι να συμμετέχουν στις εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αρκετά σοβαρή αξιολόγηση, αυστηρή, ενδημοσιάστηκα από αυτά που είπε η κυρία Ρένα από τη Δανία όσον αφορά την απόφαση για το TV2 και είναι σοφές μήνυμα για όλους μας αυτό ότι δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να αλλάζουμε τον νόμο όπως με διαφορετικό τρόπο, κάτι που εξήγησε το δικαστήριο. Το ερώτημά μου αφορά την εκ των προτέρων αξιολόγηση. Και το θέτω αυτό σε όλα τα μέρη του πάνελ. Αυτή εκ των προτέρων αξιολόγηση πώς μπορεί να εφαρμοστεί με έναν τρόπο που δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη. Διότι βλέπω αρκετές άλλες υποθέσεις περί ανταγωνισμού ή κρατικών χορηγήσεων ότι αν πρέπει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη προσέχουν ιδιαίτερος. Κινούνται σε περιορισμένα περιθώρια. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την απόφαση TV2. Και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του, άκουσα και αυτά που είπε η SET, που εκπροσωπεί τον ιδιωτικό φορέα, ότι υπάρχει περιθώριο κάτι μέλη με την αξιολόγηση των προτέρων. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Τα κράτη-μέλη θα είναι πολύ περιοριστικά. Πώς μπορεί να εισαχθεί αυτό το μέτρο αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώριο για το, να κινηθούν καλύτερα στο μέλλον οι δημόσιοι φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπαντία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία αυτή να οργανώσουμε αυτήν την ακρόαση και να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό και τώρα στο τέλος αυτής της ακρόασης βλέπω ότι ήταν πάρα πολύ θετικές ε, όλες οι ομιλίες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρεμβάντες. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σχέση με την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Θεωρώ ότι είναι θετική η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας την οποία πήρε την πρωτοβουλία να κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή, διότι πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο γίνει η αναπροσαρμογή του περιεχομένου τη αρχή του 2001 σε κάποιε αλλαγέ. Υπάρχουν αλλαγές στον τεχνολογικό τομέα, και, καθώς και στις, ε, στην νομοθεσία. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή ποιος είναι ο τόσο σημαντικός ρόλος των ε, κρατικής αυτής υπηρεσίας στα πλαίσια της δημοκρατίας και του πλουραλισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε μία ισορροπία ώστε κάποιοι με δημόσιους πόρους να μην προσετεριστούν όλη την αγορά. Είναι σημαντική η αρχή της Επικουργότητας και αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή μας σε θέματα τέτοιου μην διαδραματίζει ρόλο πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να πω ότι η, τα δημόσια κανάλια με κρατικές ενισχύσεις και με άλλες ενισχύσεις είναι και ανταγωνιστικές στον τομέα των διαφημίσεων. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούν να έχουν καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προγράμματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σαφέστατο και ενισχυμένο νομοθετικό πλαίσιο που να αφορά την παροχή υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Πιστεύω επίσης πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την δυνατότητα κάποιες ε, υπηρεσίες που παρέχονται από τις, τα δημόσια οπτικοακουστικά μέτρα να πληρώνονται κατά κάποιο τρόπο από τους πολίτες. Βεβαίως, η δημόσια, οι δημόσιες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέτρων ξέρουμε ότι είναι δωρεάν για τους πολίτες, δεδομένου ότι πληρώνονται υπηρεσία αυτή με άλλο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους για τη συνεισφορά τους που ήταν εξαιρετικής ποιότητας. οι παρατηρήσεις τη συναδέλφου Ιερώνημη θα πρέπει να μπουν στα πρακτικά της συνεδρίασης. Και πιστεύουμε ότι πρέπει οι γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν που έχουν σχέση με αυτό το θέμα να συνεργαστούν με μας. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό που δεν είναι παρούσα η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε αυτό να το κολυσορίσουμε και να περιμένουμε ε, ε, να υπάρχει και θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρχει μια συνεργασία προς όφελος των ευρωπαϊκών συμφερόντων όταν αναφερόμαστε ποια εικόνα θα πρέπει να έχουν τα ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει η λογική του δικαίου του ανταγωνισμού αφενός και της πολιτισμικής ε, πολυμορφίας πλουραλισμός των ΜΜΕ και ποιοτικό περιεχόμενο αυτά θα πρέπει να είναι σε ισορροπία και δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε τα πράγματα στα χέρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Κατόπιν θα ήθελα να τονίσω ότι παρά είναι πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει ένας καλός αναγνωσμός μεταξύ των εκπροσώπων του ιδιωτικού και δημοσίου ε, τομέα. Έχω μια ερώτηση προς τον Ρος Από ό,τι σας κατάλαβα, θεωρώ ότι η προτάση Σαρκοζή να μην υπάρχει ε, καμία διαφήμιση στους ε, δημόσιους φορείς σας φαίνεται καλή. Και μετά θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση προς τον κύριο Πράγμα. Είπατε ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός είναι Google, Google, Facebook και οι διάφορες υπηρεσίες ίντερνετ. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται στο μέλλον όταν πρόκειται για πολιτικές λύσεις. Προς τα πού θα κατευθυνόστε εσείς. Ποιοι είναι οι διαγωνισμοί που θα πρέπει να έχουμε κατά νου εν ώψη αυτών των μεγάλων παικτών που άλλαξαν τόσο πολύ την εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πριν δώσω ε, το λόγο για πέντε λεπτά, ε, για πέντε λεπτά σε όλους τους ε, εισηγητές και θα ήθελα να αρχίσω από το τέλος προς την αρχή. θα ήθελα δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις περισσότερο... καταρχήν, πριν κάνω τις δύο ερωτήσεις, είναι, θα ήθελε η Κομισιόν να πάρει το... Α, sorry. Ναι, δύο λάθη. Η κυρία ε, Τομαζεύσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να πω κάποια πράγματα, μερικά λόγια σχετικά με το θέμα που κουβεντιάζουμε. Αφού έχω την ευκαιρία λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι το πρώτο πρόβλημα είναι σαφείς δημοσιονομικοί κανονισμοί, κανόνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να αναφερθώ στη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στην Πολωνία όσον αφορά τις εισφορές για τη συνδρομή, για την άδεια. Γιατί η κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην Πολωνία από τι άδειε ε, χρηματοδοτούνται, από την συνεισφορά του θεατού και του ακροατού δηλαδή. Και θα ήθελε να απαλλαγεί αυτό το σύστημα η κυβέρνηση από την άδεια. Όμω, οι εκπρόσωποι των μέσων και διάφοροι άλλοι φορεί εμπλεκόμενοι υπερασπίζονται αυτή την άδεια για τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αυτή την εισφορά. Διότι έτσι παρέχεται κρατική ενίσχυση. Αλλά δεν είναι άμεση επιχορήγηση κρατική, τι ο τρόπος είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των κρατικών φορέων και των μέσων ενημέρωση. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι έτσι μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με ένα δημοκρατικό τρόπο. Να παίζει δηλαδή το ρόλο της το σωστό η κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο ανεξάρτητα από το ποιος έχει την εξουσία, ποιος είναι στην κυβέρνηση. Και θα σας πω ότι αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα στην Πολωνία. Για ένα χρόνο τώρα. Ξεκίνησε και κατά ένα χρόνο αυτή η συζήτηση. Θα πρέπει ίσως να μιλήσουμε διάφορες μορφές κρατικών ενισχύσεων και επιχορηγήσεων. Πρέπει, μάλλον σαν ερώτημα το θέτω αυτό. Πρέπει να συζητούμε διάφορε μορφέ κρατική ενίσχυση. Δεύτερον, διαφημίσει. Ε, έχουμε ένα μεικτό σύστημα κι εμεί. Ο βαθμός όμως, ε, το ποσοστό των διαφημίσεων είναι χαμηλό ε, στα κρατικά κανάλια. Τα προγράμματα, παραδείγματο χάρη, δεν μπορούν να διακοπούν για να μεταδοθούν διαφημίσεις στην τηλεόραση και υπάρχουν και περιορισμοί όσον αφορά ε, και το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τα προγράμματα τα οποία μπορούν να εκπέμπονται συγκεκριμένες, σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες, ορισμένες ώρες. Τώρα, όσον αφορά κάτι που είπε η κυρία Χένικοτ Νομίζω ότι η άποψή της σχετικά με την ποιότητα της κρατικής τηλεόρασης των κρατικών μέσων είναι πολύ σημαντικό θέμα στην Πολωνία. Ένα πρόγραμμα, το Big Brother, είναι πολύ δημοφιλές στην Πολωνία, συγκεκριμένη ώρα. Ήταν μάλλον μια συγκεκριμένη περίοδο πολύ δημοφιλές το Big Brother. Και κάποιος από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εξελέγει βουλευτής στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Ε, είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας, να το θυμόμαστε. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας δηλαδή ότι καμιά φορά τέτοια προγράμματα μπορούν να έχουν και κάποια επιρροή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνάδελφο. Μήπως θέλει να πάρει το λόγο κάποιος από την Επιτροπή, ε, από τη Διεύθυνση Πληροφόρησης, Κοινωνίας Πληροφόρησης, είναι εδώ. Ε, θα ήθελα πριν δώσω το λόγο για τρία λεπτά στους ε, προσκεκλημένους μας. δύο συμπληρωματικά ερωτήματα, αυτών των οποίων έθεσα στον καθένα ξεχωριστά. Ε, θα ήθελα, ε, αν είναι δυνατόν, να μας πείτε σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευση και η εξέλιξη της κατανομής του ψηφιακού μερίσματος και των ε, συχνοτήτων μετά από τις πρόσφατες αποφάσεις έτσι ώστε για να δούμε το θέμα και της πρόσβασης των τηλεπικοινωνιών στο χώρο του ψηφιακού μερίσματος πώς πηγαίνει αντίστοιχα, ένα. Ε, και το δεύτερο, ε, μία ερώτηση ε, σχετικά με, το, την... στο Ζαπιό, κύριο... Το είπα καλά. Σχετικά με το θέμα της evaluation των προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης τα οποία με βάση αυτή την αξιολόγηση θα γίνεται και η ενίσχυση ή ο βαθμός ενίσχυσης, αν το κατάλαβα καλά, της κρατικής τηλεόρασης. Θα είναι ποιοτικά, ποσοτικά τα κριτήρια, θα λαμβάνουν ε, στόχο κάποια άλλα κριτήρια τα οποία είναι εκπαιδευτικά, πολιτιστικά ή και ανταγωνιστικά σε σχέση με την ιδιωτική τηλεόραση. Ε, τόσο για το θέμα της, evaluation, ε, ε, της evaluation το οποίο ζητάει η Επιτροπή είναι σημαντικό και νομίζω ότι ο κύριος Φίσερ το έθεσε. Ε, ας αρχίσουμε με τον Πασκάλ. Τρία λεπτά ο καθένας. Τρία λεπτά. Nicht an, doch. Ja, pardon. Αναφέρθηκατε στο ψυχιακό μέρισμα. Υπήρχαν ε, κάποιες ενδείξεις ότι ορισμένοι παίκτες πραγματικά και εδώ ε, τοποθετήθηκαν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του αναγωνισμού με δύο λόγια, εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική για τις συχνότητες θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών για τον τομέα της ε, ραδιοτηλεόρασης και ότι εδώ πρόκειται για έναν τομέα όπου διαγνωσμός δεν μπορεί να θεωρηθεί αποχωρισμένος από το υπόλοιπο. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί όλους ιδιαίτερως και γι' αυτό ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την οργάνωση της ακρόσης αυτής. Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι χρειαζόμαστε αυτή τη συζήτηση και το θέμα του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού στο σύνολό του. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικό σκεπτικό στον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από σκοπιά μα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ιδέα αυτή της ουδετερότητας της τεχνολογίας να προωθηθεί με συνέπεια. Να σεβαστούμε αυτό που τα αρμόδια κράτη-μέλη θέλουν για το δημόσια ραδιοτηλεόραση. Οι συζητήσεις γίνονται κυρίως στα κράτη-μέλη. Για τους υπηκόους των οποίων, οι οποίοι πληρώνουν κιόλας, προετοιμάζονται τα προγράμματα αυτά. Είναι νομίζω σαφές για όλους ότι μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα διακονισμού, το λεγόμενο διτό σύστημα, Βέβαια υπάρχει και εδώ ισορροπημένος ανταγωνισμός, είναι σίγουρο αυτό, μαθαίνουμε εμείς από εσάς, εσείς από, από μας. Ο ανταγωνισμός παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το ανέφερα και εγώ και άλλοι. Δεν πρέπει δηλαδή να χάσουμε το στόχο από τα μάτια μας γιατί εδώ πρόκειται για το θέμα της ευρωπαϊκής παρουσίας σε ένα διεθνές δίκτυο στο οποίο υπάρχουν ε, συμφέροντα πέρα από το οικονομικό. Γιατί εδώ προωθούνται οι πολίτες προς ένα συγκεκριμένο ε, περιεχόμενο. και πρέπει οπωσδήποτε να εξακολουθεί να είναι παρούσα η Ευρώπη και εδώ. Και μου φαίνεται τελικά πολύ σημαντικό μια που η βάση μας είναι ανταγωνισμός και οικονομία οι θετικές επιπτώσεις των δημοσίων επενδύσεων στον τομέα αυτό θα πρέπει να αναγνωριστούν. Αναγνωρίζονται Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όμως πιο σαφέστερα όταν εφαρμοστεί στην πράξη αυτό. Γιατί ο οικονομικός μας ρόλος δεν πρέπει να θεωρηθεί πάντα αρνητικά σαν ε, έναν στρεβλωμένο ανταγωνισμό. Η ΕΤΕΦ θα επενδύσει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη χρονιά και ελέγχει πόσο πιο μεγάλο σημαντικό ρόλο παίζει αυτό σε μικρές χώρες. Αξίζουμε τα χρήματά μας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ευχαριστώ, ο κύριος το λόγο. Εκτός μικροφώνου, κύριε Βράβετς. Α, ναι, εντάξει τώρα. Τρεις ερωτήσεις υπήρξαν το πρώτο, η διαφήμιση στους δημόσιες ε, υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό στο μέλλον να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να ε, χρηματοδοτούνται στο μέλλον οι υπηρεσίες αυτές και μέσω διαφήμιση γιατί αυτό παίζει ειδικό ρόλο στις μικρές αγορές. Ε, δεύτερο, η προστιθέμενη αξία που δημιουργούν. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Υπάρχουν, υπάρχουν ε, ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και θα πρέπει εμείς ε, ως δημόσιες υπηρεσίες να αντιμετωπίσουμε τις συζητήσεις αυτές και θα πρέπει να φροντίσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά τα ποιοτικά κριτήρια. Ποσοτικά κριτήρια είναι σχετικά απλά για να κοιτάξουμε παραδείγματο χάρη πόσοι εκπρόσωποι υπάρχουν εδώ από δημόσιες υπηρεσίες στο, στις Βρυξέλλες και πόσοι είναι οι φίλοι μας από τους εμπορικούς ε, υπηρεσίες. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά όσον αφορά και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Και τέλος την ερώτηση της κυρίας Τρούπελ. Είναι τεράστια ε, πρόκληση. Ε, αυτό που κάνει η Google ε, με διαφήμιση στο λεγόμενο behavioral targeting. Να κοιτάνε δηλαδή τι ενδιαφέρει τον κάθε ένα πολίτη. Στην Αυστρία το 15% της διαφήμισης γίνεται μέσα στα πλαίσια των ε, προγραμμάτων mail, των ε, μηχανών αναζητήσεων ε, κλπ. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα αλλάξει η μορφή και για τις δημόσιες υπηρεσίες της δηλαδή τηλεόρασης και για τις ιδιωτικές και θα πρέπει να δούμε πού δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά στα ΜΜΕ και πού θα πρέπει τα ΜΜΕ αυτό που είναι ένας ακρογωνίος λίθος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας να χρηματοδοτείται στο τέλος. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό ερώτημα για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δίνω το λόγο στην Μαρία Ραν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα που με απευθύνθηκε και γι' αυτό θα ήθελα να εστιαστώ στην εκ των προτέρων αξιολόγηση, εξάντε αξιολόγηση. Όπως προβλέπεται στο σχέδιο ανακοινώσεως τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν αφορά μόνο την κατάχρηση, αλλά αφορά τη γενική διαδικασία για το δημόσιο φορέα. Τι θα πρέπει να κάνει το ξεκινά μια νέα υπηρεσία ή αν επεκτείνει η φυστάμενη υπηρεσία. αναφέρει ξεκάθαρα στην ανακοίνωση ότι όσο πιο κοντινή είναι η νέα υπηρεσία στις φυστάμενες εμπορικές υπηρεσίες είναι πιο πιθανό να απομακρύνει τους θεατές από τους εμπορικούς φορείς και θα στρεβλώσει και να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Αυτό σημαίνει ότι όποτε ένας δημόσιος φορέας θέλει να ξεκινήσει μια νέα υπηρεσία θα στρεβλώνει τον ανταγωνισμό εκτός εάν δεν έχει εμπορική δυνατότητα, εμπορικό, εμπορική προπτική αυτή η υπηρεσία ή δεν προσφέρεται από έναν άλλο φορέα στην αγορά καθόλου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους δημόσιους φορείς, διότι παρεμποδίζει την ανάπτυξη του δημόσιου τομέα, του δημόσιου φορέα και των υπηρεσιών που παρέχονται. De facto, ο ιδιωτικό φορέας, ο εμπορικός φορέας θα είναι εκείνος που θα επηρεάζει το τι θα κάνει στο μέλλον ο δημόσιος φορέας. Το είδαμε ήδη αυτό στις συζητήσεις που είχαμε με, τους, με τον τομέα των εφημερίδων. Ότι ξεκινήσαμε στη Δανία στο διαδίκτυο, τη χρήση του διαδικτύου εδώ και 15 χρόνια. Και τώρα που υπάρχουν δυνατότητες στην αγορά και υπάρχει περιθώριο διαφημίσεων στο διαδίκτυο, θέλουν να μας βγάλουν από το διαδίκτυο εμάς. Γι' αυτό το θέτω έτσι το θέμα, ότι θα πρέπει εδώ η αρμοδιότητα συνδέεται με το τι κάνουν οι ιδιωτικοί φορείς. Και είναι τεράστιο και το ε, γραφειοκρατικό άχθος. Αυτή η αξιολόγηση που απαιτείται είναι τεράστιο το βάρος. Είμαστε μικρή χώρα, έχουμε πολύ χαμηλότερο προπολογισμό σε συγκρίση με τι μεγαλύτερες χώρες στην Ευρώπη. Έτσι, εμποδίζεται η κανονική ούτως υπήν ανάπτυξή μα. Γιατί ε, δεν μπορούμε να παράγουμε τόσο περιεχόμενο που θα έχουμε λιγότερο χρήμα στη διάθεσή μα. Αυτό μα ανησυχεί πάρα πολύ και το θεωρούμε το σημαντικότερο ζήτημα. Δεν θέλουμε να γίνεται γενική ευρωπαϊκή εξάντε αξιολόγηση, των τροπών αξιολόγηση. Ο εθνικό νομοθέτη θα πρέπει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρία. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Μπίγκαμ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. τρία ερωτήματα πρέπει να απαντήσω. Το πρώτο ήταν δικό σας και της κυρίας Ιερώνημη. Δηλαδή, κατά πόσο η κοινωνία των, ε, της πληροφορικής, των πληροφοριών που συνδέεται, συνδέεται με την επικοινωνία, με την ανακοίνωση, συγγνώμη. Δεν θα πω εγώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι να κάνει, μακάρι να μπορούσα. Και όσο αξίζει η άποψή μας, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Αν υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση και όχι απλώς ένα κείμενο της Γενικής Διευθύνσης περί ανταγωνισμού. Το δεύτερο ερώτημα, αυτή η κυρία Τρίπελ, για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Γαλλία, όπου ο εκεί έχει πολύ πιο περιορισμένες δυνατότητες διαφημιστικές. Και πρόθεση είναι όταν γίνει η ψηφιακή αλλαγή, πάψουν οι αναλογίες εκπομπές να είναι μηδέν οι διαφημίσεις. Ε, είπατε ότι φαντάζεστε ότι αυτό το θεωρώ καλό. Είναι σημαντικό να κάνουμε διαφοροποίηση εδώ. Η αρχή, σύμφωνα με την οποία να παίρνουν δημόσιους πόρους και μόνο οι δημόσιοι πάροχοι, είναι σωστή Σωστή η ιδέα. Όμω το πώ εφαρμόζεται αυτό στη Γαλλία έχει πολύ σοβαρέ συνέπειε για τον ειδικό τομέα. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται για κάθε χώρα από τα 27 κράτη. Ο συνάδελφο του TFAN έφτιαξε ένα πολύ μεγάλο έγγραφο που είναι διαθέσιμο στο βάθο τη αίθουσα. Και η CSR θα αναφερθεί στο θέμα μετά από μένα. Ποιο είναι το πρόβλημα με το γαλλικό σύστημα. Αντί να, να αντικαταστήσουν αυτό που χάνουν από τι διαφημίσει με δημόσια χρήματα, επιβάλλεται ένα φόρο στους ε, δημόσιους φορείς και θεωρούν ότι θα γίνει η ροή των χρημάτων από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό. Τι συμβαίνει, η διαφήμιση πήγε αλλού, άλλαξε χέρια, πήγε στο διαδίκτυο, πήγε στον έντυπο τύπο ή αλλού. Οι Γάλλοι δημόσιοι φορείς πληρώνουν αυξημένο φόρο με μειωμένα έσοδα. Καλύτερα διαβάστε το. Διαβάστε το, μην ακούτε τι λέω εγώ, ποια ερμηνεία δίνω. Ο κ. Φίσερ έθεσε ένα ερώτημα για τον εκ των προτέρων, αξιολόγηση. Θα ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό, τι συζητάμε. Η ECT και εγώ δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Οι δημόσιοι φορείς να χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία. Το να, μαραίνον να μαραίνονται οι δημόσιοι φορείς σε αναλογικό χώρο ενώ όλα γίνονται ψηφιακά, αυτό είναι φαντασίες, εφάνταστα πράγματα μπορούν να έχουν και ψηφιακά κανάλια, δημόσιοι φορεί και online υπηρεσίε. Το θέμα είναι πώ τα ρυθμίζεται ο νέο κόσμο. Και πού διαφωνώ με τη γειτόνισά μου από τη Δανία είναι το θέμα τη λεπτομέρεια στην επικοινωνία. Το σχέδιο, επικοινωνία, το σχέδιο ανακοινώσεω, συγγνώμη, έχει ακριβώ 9 παραγράφου όσον αφορά τον εκ των προτέρων έλεγχο. Οι τρει πρώτε παράγραφοι αναφέρονται στι αρμοδίε των κρατών μελών και στην παράγραφο 62 αναφέρονται ιδιαίτερε περιστάσει όταν τα κράτη-μέλη δεν έχουν ανεξάρτητο ελεκτικό ρυθμιστικό φορέα. Η λεπτομέρεια ρυθμίζεται στο εθνικό επίπεδο. Στο Ενωμένο Βασίλειο η συμφωνία μεταξύ BBC Trust και Ofcom ε, είναι μια συμφωνία 36 σελίδων. Στη Γερμανία Συμβασμό Εξωτερική Επιτροπή και των Ομοσπονδών Κατηδίων είναι 90 σελίδε έγγραφο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα έδωσε 9 παραγράφου γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει τι γενικέ αρχέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σωστό αυτό. Και η λεπτομέρεια πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Και αν είσαι μικρότερο κράτο μέλο, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο λεπτομερή όσο η Ofcom και οι γερμανικέ ρυθμιστικέ αρχέ. Αν μπορεί να περιγραφεί η κατάσταση στη Γερμανία σε έξι σελίδε, δεν έχουμε πρόβλημα. Δύο από του τρει δημόσιου φορεί που μίλησαν από τη Γερμανία και τη Δανία ήταν ενδιαφέρον να δούμε ότι ήδη έχουν συστήματα εκ των προτέρων αξιολόγηση. Το θέμα είναι να σταθμίσουμε τα πράγματα. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία μια νέα προσπάθεια σε σχέση με τι συνέπειε που έχει αυτή η νέα προσπάθεια για την αγορά. Ευχαριστώ, Ε, το λόγο στον κύριο Ζαπιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να απαντήσω το δικό σα ερώτημα πρώτα απ' όλα για την εξάντε αξιολόγηση των εκπομπών των ε, κρατικών. Αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως ήταν μια πρόταση του κυρίου Μπουγιό, πρόεδρου του Συμβουλίου του Οπτικοακουστικού Συστήματος, την οποία δεν ακολούθησε η γαλλική κυβέρνηση. Η ιδέα του είναι να έχουμε μία ένα πίνακα αξιολόγηση, μια κλίμακα αξιολόγηση όπως είπα όλων των εκπομπών και να τις βαθμολογήσουμε με βάση ένα ποιοτικό κριτήριο και να δούμε γιατί μια τέτοια εκπομπή καλύτερα να μεταδίδεται από την κρατική τηλεόραση παρά από ένα ιδιωτικό κανάλι. Βεβαίω τι ενδιαφέρει τα κανάλια το ποσοστό τηλεθέασης, ενώ το κρατικό η ποιότητα, διότι έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Τώρα για να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Ιεχονιμή. για τα διάφορα προγράμματα αλλά la carte, όπως λέγαμε. Ο νόμος περί οπτικοοξικών μέσων θα, όπως σας είπα, θα δημοσιευθεί έως το τέλος της εβδομάδας και η υπεύθυνη ανεξάρτητη αρχή οπτικοοκουστικών μέσων θα πρέπει να ρυθμίσει μια τέτοιου είδους ε, ε, υπηρεσία. Δηλαδή προγράμματα τηλεόρασης ή βίντεο à la carte. Λαμβάνοντας υπόψη πώς θα ρυθμιστεί η διαφήμιση, ποιες ε, παραγωγές πρωτότυπες γαλλικές ή ευρωπαϊκές θα και τρίτον πώς θα προστατευτούν τα παιδιά. Αυτό ζητείται από την ανεξάρτητη αρχή να λάβει υπόψη και να ρυθμίσει και βεβαίω τα διάφορα θέματα δεντολογής. Τώρα, οποιαδήποτε άλλο θέμα συμβάσεων, τιμών, ε, είναι θέματα που αφορούν τα διοικητικά δικαστήρια. Ή τον νόμο που ισχύει και για τα άλλα θέματα. Αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, τώρα θα ήθελα σε σχέση με αυτό το που ο κύριος Μπίγκαμ για το θέμα των φόρων να πω το εξή. Στι διάφορε κοινοβουλευτικέ συζητήσει που έγιναν, είπαμε ότι δεν πρόκειται για ποσά τα οποία πηγαίνουν απευθεία στην τηλεόραση. Είναι ποσά τα οποία προέρχονται, λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια του ε, κρατικού προϋπολογισμού και μετά δίδονται στους διαφόρους. όταν τα δικαιούνται. η κυβέρνηση, ίσως όχι λόγω της οικονομικής κρίσης του 2009, αλλά τα επόμενα χρόνια πιστεύει ότι θα πρέπει ένα μέρος των ε, κερδών της διαφήμισης να πάει και στα ιδιωτικά κανάλια. Και βέβαια όλα είναι αναλογικά ανάλογα με τον τζίρο που κάνει το κάθε κανάλι. Θα είναι μικρά τα ποσά, αλλά πρέπει να σας πω ότι νομικής απόψεως δεν πρόκειται για ποσά τα οποία δίδονται για τα δημόσια οπτικοακουστικά μέτρα. Και τελειώνοντας, θα πρέπει να πω ότι χαίρομαι διότι πολλοί τόνισαν τη σημασία της αρχής της ε, επικουρικότητας της ανακοίνωσης της Επιτροπής και την ανάγκη για την δημόσια αυτή υπηρεσία να μπορέσει να στραφεί στο μέλλον και να ανταποκριθεί σε σχέση με την ψηφιακή τηλεόραση στις προσδοκίες των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ε, δίνω το λόγο στον ε, κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε δύο θέματα από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, όλοι, πολλοί από εμά αναφερθήκαμε στο γαλλικό ε, σύστημα, τα νέα κριτήρια χρηματοδότησης. Πρέπει να σας πω ότι εμένα καταρχήν καλό μου φαίνεται αυτό. Δηλαδή, οι ιδιωτικές τηλεοράσεις όσο ελευθερώνουν τα κρατικά κανάλια ζώνες διαφήμισης, θα πρέπει να μπορούν εκείνοι να την πληρώνουν. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα θα πει είναι ένας ε, τρόπος ο οποίος να υποχρεώνει όλους να βρίσκουν χρήματα διαφημίσεις με τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα με τις ε, ε, παραδόσεις, με τις συνήθειες, με τις δυνατότητες, ο καθένας θα πρέπει να προσπαθεί να βρει έναν τρόπο με τον οποίο να εφαρμόσει αυτή την αρχή, που μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα στο σέρις. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο ελέγχθη προηγουμένως, η σύγκληση των μέσων όπως έλεγε και η Επίτροπος Ρέντιν, να κάνουμε αυτό προγραμματισμό κατά κάποιο τρόπο. Ο εκπρόσωπος της ΟΕΡΤΕΦ είπε τι σημαίνει αυτό για τον ανταγωνισμό. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια δυνατότητα που δίδεται στις δημόσιες τηλεοράσεις. Αυτή η σύγκληση μέσων όπου η... το ίντερνετ είναι πάρα πολύ σημαντικό πρέπει να μας βοηθήσει στο εξής. Δίδεται μία δυνατότητα περαιτέρω πληροφόρησης, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα σύν για την δημόσια τηλεόραση, για τα δημόσια κανάλια. Επίσης, όπως είπε και η Δανία εκπρόσωπα, πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα γραπτά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, καταλαβαίνω ότι η δημόσια τηλεόραση θα μπορούσε να προσφέρει από τα προγράμματα τα οποία μπορεί να κατεβάσει από το ίντερνετ ε, από αυτά τα προγράμματα να μπορέσει ε, να δώσει κάποια χρήματα ώστε να μπορεί κανείς να έχει τη δυνατότητα να κατεβάζει τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και ε, χωρίς να είμαι λόγω θέσης να μπορώ να πάρω μια προσωπική θέση ως πρόεδρος της Επιτροπής, μόνο ένα προβληματισμό θέτω στους ηθήνοντες των οπτικοακουστικών μέσων, ότι η κατάργηση της διαφήμισης, και δεν μιλάω για κατάχρηση της διαφήμισης στο δημόσιο τομέα, και η χρηματοδότηση της ε, κρατικής τηλεόρασης μόνο από δημόσιους πόρους εξαρτάται και από το μέγεθος και από τη δυνατότητα κάλυψης του δημόσιου προπολογισμού ενός μέσου πολιτιστικού χαρακτήρα πολυγλωσσίας. Αυτό λοιπόν ας το θέσουμε στα υπόψη μας, διότι δεν είναι σκόπιμο να έχουμε δύο ταχύτητες του μέσου επικοινωνίας πολιτιστικού διαλόγου εκπαίδευσης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις προτεραιότητες του κάθε εθνικού προπολογισμού. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Θεωρώ με την παρουσία ή χωρίς την παρουσία της Επιτροπής ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ως πολιτική μπήκαμε στα βαθιά του κόσμου των ακουστικών, όπου όσο μπαίνουμε τόσο πιο ενδιαφέρον είναι. Έχετε πολλά μυστικά, πολλές προκλήσεις, πολύ ενδιαφέροντα. Ε, και νομίζω ότι αυτή η audition θα ξαναγίνει ε, σε συνεργασία με την ΕΚΟΝ και την Ήτρε στα πλαίσια της συζήτησης για τις κρατικές ενισχύσεις στον οπτικοακουστικό τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, τους διερμηνείς, εσάς, τους συναδέλφους και τους βουλευτές. Καλό απόγευμα.